και καλωσορίσατε σε αυτή την απογευματινή συνάντηση. Θα είμαι ο συντονιστής, θα μιλήσω γαλλικά, γι' αυτό όσοι δεν καταλαβαίνουν γαλλικά παρακαλούνται να βάλουν τα ακουστικά τους. Σήμερα το απόγευμα έχουμε ένα πολιτικό πάνελ δεδομένου ότι έχουμε μαζί μας τους ευρωβουλευτές που είναι υπεύθυνοι για τους διάφορους φακέλους. Έχουμε τρεις εισηγητές και τρεις συντονιστές. Ελπίζω ότι σήμερα το πρωί σας εξήγησαν τι είναι, ποιος είναι ο εισηγητής, ποιος είναι ο συντονιστής. Οι συντονιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο καθένας, δεδομένου ότι, για να το συντομεύσω, είναι αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται τις διάφορες εκθέσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξ ονόματος της πολιτικής τους ομάδας και οι συντονιστές είναι αυτοί οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ηγούνται των διαπραγματεύσεων για να υπάρξουν οι συνενέσεις και οι συμβιβασμοί για τις διάφορες εκθέσεις τις οποίες συντονίζουν. Σε γενικέ γραμμέ. αυτά. Και βεβαίως ο ίδιο ο εισηγητή έχει την δική του ευθύνη, δεδομένου ότι είναι εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει την έκθεση να την παρουσιάσει ε, εξ τη της ε, Επιτροπής του στην Ολομέλεια όπου θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί. Εξ ονόματος, λοιπόν των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Μασίπη μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Νομικής Επιτροπής. Ο κύριος Μασίπη είναι μέλος Επιτροπής των υποθέσεων, αναπληρωτής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Σας εξήγησαν τι είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σήμερα το πρωί. Ιστορικές υποθέσεις, πολιτικές ελευθερίες και δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια κοινοβουλευτική επιτροπή με μεγάλο γόητρο και μέχρι πριν από λίγα λόγια Πρόεδρο τη ήταν, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, πρόεδρο τη Ιταλική Δημοκρατία, ο κ. Ναπολιτάνο. Ο κ. Μασίπη Δάλγο είναι δικηγόρος, σπούδασε νομικά. Βουλευτή από το 1972, δήμαρχος του Οβιέδο, στην περιοχή Αστούριας, στο παρελθόν. και βεβαίω, είναι μέρο του σοσιαλιστικού κόμματο ε, της Ισπανίας, ήταν πρόεδρο του Ινστιτούτου στις Αστούριες, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 και έχει διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στο κόμμα του, στην Ισπανία. Η κυρία Βίξτρομ. είναι μέλος του πάνελ, είναι μέλος των, της ομάδας των φιλελευθέρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Βίλκστρομ είναι από την Σουηδία, είναι μέλος της, Επιτροπής, ε, της Νομικής Επιτροπής και της ΛΥΜΠΕ. Έχετε σπουδάσει θεολογία στην Σουηδία και είστε, είσαστε και υπουργός ε, για 8 χρόνια των εκκλησιών στη Σουηδία. Και είναι τώρα η πρώτη σας θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξελέγει το 2009. Είσαι επίσης μέλος του Σβουλής της Σουηδίας. Και αν κατάλαβα καλά, Από το 2002 είστε μέλος της Εθνικής Επιτροπής της Σουηδίας για την UNESCO. Ξέχασα να αναφέρω ότι ο κύριος Ιδάλγο είναι εισηγητής για τα θέματα που αφορούν τις μίνιμουμ προδιαγραφές για την υποδοχή των ετούντων. η κυρία Βίλστρομ για την ε, κανονισμό του Βλίνου. ο κύριος Ρούιτο Βάρε, είναι μέλος της, των Πρασίμων. Έχουμε και μετάφραση από πρωτοελικά. Βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα. Είναι αντιπρόεδρος της ε, ειδική Επιτροπής το οργανωμένο έγκλημα τη διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, καθηγητής και συγγραφέας διαφόρων βιβλίων. Και euh, euh, η έκθεσή του, η έκθεση την οποία είναι εισηγητής, αφορά το κοινό, ε, κοινοτικό πρόγραμμα για θέματα μετεγκατάστασης και μετακίνησης. Ο κύριος Κίρκοπ είναι επίσης αντιπρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, την ε, διαφθορά και το ξέπλυμα δομικού χρήματος, μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1999. μέλος της ομάδας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, όπου στην ομάδα αυτή έχουμε κυρίως Βρετανούς συντηρητικούς, Πολωνούς και Τσέχους. Ο κύριος Κίρχοπ είναι δικηγόρος επίσης από το 99 πρόεδρος των συντηρητικών φίλων του Ισραήλ ε, αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών ε, από το 95 μέχρι το 97 για διάφορα θέματα που αφορούσαν την ε, μετανάστευση, την ε, αδειοδότηση και το παιχνίδι, την διεθνή αστυνομική συνεργασία κτλ. Ο κύριος Μάριο Μπουργκέτσιο είναι μέλο της Λίγας του Βορρά. Είναι εδώ εξ ονόματος ε, της ομάδας της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Μέλος ε, της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών επίσης. Είναι επίσης και μέλος της Ειδικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα, τη Διαφθορά και την Νομιμοποίηση Παρανόμων Εσόδων και είναι φυσικά και νομικός από το 1977 ήταν πρόεδρος της κυβέρνησης της Παντάνια από το 1994 στο 2004, πρόεδρος της ε, Λίγας του Βορρά στο Πιεδεμόντιο και μέλος ε, του Δημοτικού Συμβουλίου του Τουρίνο και ε, βουλευτής της Ιταλικής κυβέρνησης και έχει διατελέσει και υφυπουργός δικαιοσύνης. Ε, είναι συντονιστή στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για ε, την ομάδα της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν και τέλος ε, τον Κύπριο Ευρωβουλευτή μας, ο οποίος είναι συντονιστής εξ ονόματος της ομάδας Ενωτικής Αριστεράς, τον κύριο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη. Υποθέτω ότι θα επιστρέψει κάπου χρειάστηκε να πάει. Νάτος. We shall Είστε εδώ εκ μέρους της Κύπρου. Ο κύριος Κυριάκος Τριανταφυλλίδης είναι αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη. Σημαντικός ε, ρόλος. Είναι επίσης και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ευθεριών. Είναι εδώ στην πρώτη του... Α, συγγνώμη, διορθώνει ο μιλητής. Έχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Ζηλανδίας. Of English and Social Studies in New Zealand as well. Ε, από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ε, έχει επίσης αναπληρωτής ε, αξιωματούχος ε, για θέματα μετανάστευσης πριν γίνει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε αρκετές επιτροπές και ε, είναι και συντονιστής ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, εξ ονόματος της Ομάδας Ενωτικής Αριστεράς. Κύριε Μασίπιν Θέλετε να κάνετε μια εισαγωγή στη συζήτηση, σας παρακαλώ, για να ξεκινήσουμε, για να ακούσουμε την άποψή σας και φυσικά την άποψη της πολιτικής σας ομάδας. Καλησπέρα σας. Σας είπανε τα διαπιστευτήριά μου, την ε, ε, επαγγελματική μου καριέρα, σε περίληψη φυσικά. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω ευθύς εξ αρχής γιατί έχω έρθει εδώ. Διότι είμαι εισηγητής ε, για την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής του ασύλου. Όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής σας εδώ είμαι νομικός και επειδή έχω ζήσει στην Ισπανία στη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, ασχολήθηκα με τις υποθέσεις όχι μόνο των προσφύγων, διότι δεν είχαμε πρόσφυγες στην Ισπανία, δεν ήταν χώρα ασύλου τότε, τότε η Ισπανία, αλλά ασχολήθηκα με ε, εργατικά προβλήματα και πολιτικά ε, ζητήματα και πολιτικών κρατουμένων. Μια μέρα λοιπόν συνέβη το εξή στην οικογένειά μου. Η αδερφή μου και ο κουνιάδος μου χρειάστηκε να φύγουν από τη χώρα. Διότι τους ε, καταδίωκε η αστυνομία του Φράγκο, χρειάστηκε να διασχίσουν τα Πυρηναία και λαφρέα να περάσουν από την Ισπανία στη Γαλλία, στη χώρα της ελευθερίας. Η αδερφή μου, έγκυος 7 μηνών, ήθελε να γεννήσει ελεύθερη στη Γαλλία ε, και εν μέσω πολύ δύσκολων συνθήκων και εγώ τους περίμενα από την άλλη μεριά των συνόρων διότι ως ε, νομικός ε, και ήμουν και κάπως γνωστός στα νιάτα μου, είχα δυνατότητα να έχω διαβατήριο και να ταξιδεύω αρκετά εύκολα. Και διαπίστωσα τότε πώς η χώρα υποδοχής, που δεν ήταν τότε της πολιτικής μου οικογένειας, έτσι, ήταν η κυβέρνηση επί Σκάρντεστεν, Στέν. υποδέχθηκε την αδερφή μου, τον κουνιάδο μου και την ανιψιά μου που γεννήθηκε λίγο μέρες αργότερα, τους δέχθηκε ως πρόσφυγες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπόρεσαν να ξαναστήσουν την επαγγελματική και ακαδηματική τους ζωή στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και αυτή η οικογένεια η οποία είχε διωχθεί για πολιτικούς λόγους, κατάφερε να ξαναστήσει τη ζωή της και όταν πέθανε ο δικτάτορας και ήρθε η ελευθερία για την Ισπανία, η οικογένεια της αδερφής μου, ο κουνιάδος μου και η ανιψιά μου μπόρεσαν και πάλι να περάσουν ελεύθερα στην Ισπανία, να μετεγκατασταθούν και σήμερα ζουν ευτυχισμένα στη χώρα μας. Εγώ λοιπόν ως Ευρωβουλευτής όταν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών τίθεται αυτό το ζήτημα και με ορίζουν εισηγητοί λοιπόν, θέλω για την Ευρώπη να είναι πραγματικά η χώρα του, η, γη του ασύλου και της ελευθερίας όπως ήταν για τους δικούς μου και αυτό επιθυμώ για όλους τους ανθρώπους ε, καλή την πίστη. Και Αντιθέτως, με λύπη μου διαπιστώνω, καταρχάς ότι η κοινή γνώμη συγχαίει τον οικονομικό μετανάστη με τον ε, πολιτικό πρόσφυγα. Πρόκειται για δύο εκδιαμέτρου διαμέτρου διαφορετικά πράγματα. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον οικονομικό μετανάστη, αλλά προσέξτε, ο άνθρωπος που διώκεται στη χώρα του, διότι προασπίζεται την ελευθερία πρέπει να μπορεί να προστατευτεί στην Ευρώπη όπως βρήκε στέγη, βρήκαν στέγη δική μου και θα πρέπει να μπορούν να βρουν στέγη και θα πρέπει να τους την προσφέρουμε. Και αυτό δεν είναι τμήμα μόνο των Ευρωπαϊκών Αρχών ε, από την ε, Γαλλική Επανάσταση και μετά, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει βούλευση και να συμπεριλαμβάνεται στα κείμενά μας. Και σας διαβεβαιώ ότι χρειάστηκε πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και καταφέραμε να εγκρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ εργάστηκα για το θέμα αυτό και ασχολούμαι με το θέμα εδώ και 7 χρόνια. Και παρόλα αυτά εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι διέξοδος προκειμένου ο σεβασμός προς τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη και διαπιστώνουν διαφορετικά πράγματα να μπορούν να προστατευτούν οι πρόσφυγε που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πάντα πρέπει να γίνεται η διάκριση. Σέβομαι απόλυτα του οικονομικού μετανάστε, βεβαίω έχω πολιτική και κοινωνική δέσμευση ενώπιόν του, αλλά εδώ μιλάμε για μία προνομιούχα κατηγορία πολιτών, ανθρώπου οι οποίοι έδωσαν μάχη για την ελευθερία και θα πρέπει να είναι σύμμαχοί μα, ώστε σε όλε τι χώρε του κόσμου να υπάρχει ελευθερία. Είναι πονίδιστο το γεγονός ότι στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αφρική όταν υπήρχαν νέοι που έδιναν μάχη για την ελευθερία, εμεί δεν τίναμε δίκονους. Επισκέφθηκα όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και διαπίστωσα όμως το πρόβλημα. Θα σταματήσω γιατί καθυστέρησα. Από εκεί και πέρα θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίξτρομ, νομίζω ότι εσείς είχατε μια διαφορετική εμπειρία που σας οδήγησε να είστε τόσο ευαίσθητοι για το θέμα των προσφύγων και τη μετανάστευση και ασχολείστε με ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, το οποίο γνωρίζουν όλοι, το σύστημα του Δουβλίνου. Παρακαλώ λοιπόν, μπορείτε να παρουσιάσετε τη θέση σας στους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα με σας και θα σας μιλήσω για την ε, εμπειρία μου. Ασχολούμαι εδώ και τρεις χρόνια με τον κανονισμό του. Ο κύριος Μασίπ άρχισε την παρέμβασή του σήμερα το απόγευμα με μια πάρα πολύ προσωπική του συγκινητική ιστορία. Ε, εγώ είμαι Σουηδή, είμαστε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ουδέτερος χώρο, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω και εγώ κάτι με προσωπική μου η ιστορία. 1994-95, όταν ήμουν ιερέας. Ήταν εποχή πολέμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θυμάστε, πάρα πολλοί έφυγαν από το Κόσοβο σε ένα χρόνο ήρθαν 82.000 άτομα από το Κωσυφοπαίδιο στη Σουηδία. Πάρα πολλοί εγκαταστάθηκαν σε μικρά χωριά όπως το Ζήμα, στον οποίο ήμουν εγώ ιερέας. Γνώρισα πολλά άτομα, τα βοήθησα και κάποιο βράδυ όταν χρειάστηκε να φροντίσω κάποιο 20-25 ετών όταν μου έδωσε την αίτηση που είχε υποβάλει είδα στην πρώτη γραμμή το όνομά του και στη δεύτερη έπρεπε να γράψει γιατί ζητούσε άσυλο. Και εκείνο το βράδυ διάβασα κάποιες λέξεις που δεν ξέχασα ποτέ. Έγραφε ε, «Εθνοτική κάθαρθης». 50 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η προσωπική μου λοιπόν αυτή η εμπειρία είναι εμπειρία που έχω από το 1995 στο μικρό αυτό χωριό. Και πιστεύω ότι ήταν τότε η τελευταία φορά, ελπίζω στη ζωή μας, που είδαμε θύματα εθνοτικής κάθαρσης που ήθελαν να καταφύγουν και να ζήσουν στην χώρα μας. Για μένα ήταν πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος και ελπίζω ότι θα ήταν η τελευταία φορά. Σύντομα θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία. Είδαμε ότι και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έκαναν αίτηση για να προσχωρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα αυτό είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή της ιστορίας της Ευρώπης. Όταν βλέπουμε πραγματικά και αισθανόμαστε πραγματικά ότι έχουμε προοδεύσει έχοντας μιλήσει τώρα σε εσά για αυτή την προσωπική μου εμπειρία, έχοντας ε, και κατά νου τη δική μου δέσμευση για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, πρέπει να πω ότι από εκείνο το βράδυ άρχισε και πραγματικά τρέμω. Όταν σκέφτομαι ως πολύ νέο άτομο τότε να διαβάζω αυτή την φράση εθνοτική κάθαρση. Από εκεί ξεκίνησε η δεσμευσή μου και πριν από τρία χρόνια κληρονόμησα από τον την πρωτά κάτοχό μου τη Ζανίν Πλάσερ που έφυγε για την Ολλανδία και είναι υπουργό δικαιοσύνη τώρα, κληρονόμησα αυτό το φάκελο του κανονισμού Δουβλίνο 2. Πρόκειται για ένα σύστημα ασύλου το οποίο άρχισε με την δήλωση της του 1991 για πρώτη φορά στην Ευρώπη αρχίσαμε να μιλούμε για κοινό σύστημα πολιτικής ασύλου στην Ευρώπη και πρόκειται για μία φιλοδοξία την οποία όλο και περισσότερο θέλουμε να ηθοποιήσουμε και υπάρχει και στο πρόγραμμα της ε, της συνδικής της χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι όλη η δουλειά που επιτελέσαμε δεν ήταν εύκολη. Αντιθέτως, την ε, στιγμή των οικονομικών ε, κρίσεων και των ε, δυσκολιών, τα κράτη-μέλη πρέπει να πω ότι έχουν μεγάλους ενδιασμούς για να, την δημιουργία αυτού του κοινού συστήματος χρήσης ασύλου με βάση την λιλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όπως σας είπα, και όπως ελέγχθη είμαι εισηγητής για την αδιατύπωση του κανονισμού Δουβλίνου και ε, εργάζομαι νυχθημερών εδώ και τρία χρόνια για να ολοκληρώσω το φάκελο. Ο φάκελος πρέπει να πω ότι είχε μπλοκαριστεί για πολλά χρόνια στο Συμβούλιο και η, στα πλαίσια της Πολωνικής Προεδρίας ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις, είδαμε μια κάποια πρόοδο και είδαμε ότι προχωρούμε βήμα προς βήμα. Το μεγάλο αμφιλεγόμενο σημείο ήταν το αίτημα της Επιτροπής καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εισαχθεί αυτός ο μηχανισμός ε, της ε, ανάκλησης του καθεστώτος όταν δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες εγγύησεις, δηλαδή την κατάσταση που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να πω ότι φοβούνταν ότι ένας τέτοιος μηχανισμός της ε, ανάκλησης του καθεστώτος μεταφοράς θα δίνανε ένα πρόσχημα στην Ελλάδα σε άλλες χώρες να μην συμπεριφερθούν σωστά. Το 2011, και σας δίδω αυτό το παράδειγμα δεδομένου ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ε, σωστή απόφαση του ε, ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, MSS κατά της Ελλάδας και του Βελγίου για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν ένας Αφγανός, ο οποίος ζητούσε άδειο, μεταφέρθηκε από το Βέλγιο στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα προηγούμενο και για να μην... Ε, και έτσι σταμάτησαν από τότε και μετά όλες οι μεταφορές ε, και ανάκληση χορήγηση του ασύλου από το ένα κράτος στο άλλο. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ασχολούνται με το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναμίες σε καταστάσεις αίτησης ε, ασύλου σε ένα πολύ αρχικό στάδιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω σε όλους τους παρόντες εδώ σήμερα ότι αυτός ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όντως θα βοηθήσει την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων όπως αυτή η που συνέβη στην Ελλάδα από το να συμβεί και σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτή η προσέγγιση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να πω ότι τελικά ε, μπόρεσε να αντιστρέψει την κατάσταση στο Συμβούλιο και έγινε αποδεκτό αυτό από τα κράτη-μέλη και προχωρήσαμε προς μια συνενετική λύση την οποία ολοκληρώσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο μετά από πολύ δύσκολους ε, διαλόγους σε τριμερές επίπεδο. Ήμουν εγώ υπεύθυνη και ξέρω περί τίνος πρόκειται. Και θα πρέπει να υπάρχει μία εποπτεία στα κράτη-μέλη, ώστε όταν υπάρχουν αδυναμίες και προβλήματα σε έγκαιρο στάδιο, να γίνεται προσπάθεια να επιλύθουν. Και βεβαίω όλα αυτά θα γίνονται και με την ε, συνδρομή τη Επιτροπή, αλλά κυρίω στα πλαίσια του γραφείου υποστήριξη που υπάρχει στη Μάλτα. Πρέπει να πω ότι έγιναν πάρα πολλέ ε, βελτιώσει. Ε, δεν έχω το χρόνο δυστυχώ για να τα απαριθμίσω όλο. Απλώ κάποιες παρατηρήσει θα κάνω. Αλλά πριν να το κάνω αυτό, επιτρέψτε μου να πω το εξή. Σε έναν ιδεατό κόσμο, σε έναν ονειρικό κόσμο, ο κανονισμός του Δουβλίνου, δεν θα, τον κανονισμό του, του Δουβλίνου, συγγνώμη, δεν θα τον χρειαζόμαστε. Αλλά τώρα αυτόν έχουμε. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο ώστε να υπάρχουν πιο ισχυρές ε, νομικού τύπου εγγυήσεις και για τους πρόσφυγες και πολύ σαφείς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη διότι έχουμε και ένα άρθρο το οποίο λέει, παραθέτω, οι ετούντες άσυλο δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε κράτες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχει κίνδυνος απανθρωπής ή αναξιοπρεπούς μεταχείρισης. Πρόκειται για άρθρο 3.2 του κανονισμού. Δεδομένου ότι πρόκειται για εξαιρετική βελτίωση. Άλλες βελτιώσεις είναι η οικογένεια, η συγγενής αν θέλετε, με την ευρύτερη έννοια. Ένα ασυνόδευτο ανήλικο παιδί μπορεί σε ένα άλλο κράτος μέλος να πάει όχι μόνο με τους γονείς του, αλλά με τους παππούδες, με άλλα αδέλφια αν έχει, με θείους, με θείες και δίδονται πιο σαφείς κανόνες και καθαρές προθεσμίες για τις ε, κρατήσεις και για τις περιπτώσεις τις οποίες κάποιος ε, εκδιώκεται και πρέπει να γυρίσει πίσω. Νομίζω ότι όλα... Αυτό που μας απασχολεί είναι κυρίως το θέμα της αλληλεγγύης για τους ετούντες αλλά κυρίως νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τον ε, φαύλο κύκλο Τη δυσπιστία μεταξύ κρατών μελών. Διότι είδαμε τα πρόσφατα χρόνια ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι πραγματικά η λέξη που μπορεί να περιγράψει τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών για το θέμα τα αυτά. Θα πρέπει αυτό τον φαύλο κύκλο να σταματήσουμε, να μπορέσουμε να συστήσουμε σχέσεις αμοιβέ εμπιστοσύνης και σήμερα, και αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα γιατί το τι χρειαζόμαστε το κοινό σύστημα χωρίς ασύλου, σήμερα υπάρχουν 10 κράτη-μέλη από τα 27 που υποδέχονται 92% των ε, ετούντων άσυλο. Πράγμα που σημαίνει ότι 17 χώρες θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα αυτό ε, το λέγω για να καταλάβετε την αναλογία και τη δυσαναλογία που υπάρχει. Βέβαια, κάθε χώρα έχει τις δυνατότητές της και μια μικρή χώρα σαν τη Μάλτα που υποδέχεται πάρα πολλούς ετούντες άσυλο δεν μπορεί να βοηθήσει όσους πολλούς όπως η Γαλλία ή η Γερμανία ή η Σουηδία. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι το δικαίωμα ασύλου είναι ένα αναφέρεται το δικαίωμα. Καλύπτεται από την σύμβαση της Γενέβης. Δεν είναι θέμα γενεοδορίας. Ο καθένας δικαιούται διεθνή προστασία και θα πρέπει να του χορηγείται. Όταν θα τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία θα αρχίσουν νέες προκλήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά σε όλες τις χώρες μέλη. Η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και θα επικουρείται και από το ε, Γραφείο Υποστήριξης Ασύλου και βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι πόσο καλή είναι στη θεωρία η νομοθεσία εάν δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά ακούμε ιστορίες όπου δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε ακόμη και τα πιο ευάλωτα άτομα. Πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης μας αποκαλύπτουν τέτοιου είδους παράξενες συγκινητικές ιστορίες ατόμων προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα και προσπαθούν και προσπαθούν πράγμα το οποίο βοήθησε ε, πολλές ιστορίες να έχουν αίσιο τέλος, όχι όμως όλες. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα τόσο ασφαλές σύστημα, ώστε κανένα άτομο να μην την χάνει κακής μεταχείρισης. Διαπιστώνω ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαι όμως πεπισμένη ότι το νέο ε, νομικό πλαίσιο θα βοηθήσει τα μάλλα τη βελτίωση κατάστασης. Αν μπορούμε λοιπόν να ανεβάσουμε τον πύχη όλοι μαζί σε όλες τις χώρες μέρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ περισσότερα άτομα με ανθρώπινο τρόπο, με τον ανθρώπινο δόμο που δικαιούνται. Το να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση των συστημάτων σε ένα κοινό σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο θα αυξήσει τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα τους ανθρώπους και κανένας έτσι δεν θα μπορεί να ανεχθεί ένα, δύο ή κάποια κράτη-μέλη να μην συμπεριφέρονται σωστά ή να μην επομίζονται τις ευθύνες που έχουν. Ο κανονισμός του Δουβλίνου καθώς και η οδηγία περί υποδοχής, η για την οποία είναι ο κύριος Ιδάλγο, είναι έτοιμες για να εγκριθούν. Έχουμε ε, ε, ολοκληρώσει την περίοδο διαπραγμάτευσης. Τώρα ε, χτενίζουμε τις διαδικασίες, τελειώνουμε και ελπίζω από το βάθος της καρδιάς μου ότι θα μπορέσουμε τους φακέλους αυτούς να τους υιοθετήσουμε τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλη ευχαρίστηση αργότερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις που θα μου θέσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βίκστρομ ο κύριος Ρούι Ταβάρες. Τι θέση έχετε εσείς για το θέμα αυτό, για το θέμα των θεωρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζοντας, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω καταρχάς πορτογαλικά. Τα εθνικέ βουλέ είναι διαφορετικέ η μία από την άλλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ούτω ή άλλω διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο εθνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ήδη εσεί ε, εδώ σήμερα στην ημερίδα που είχατε, είχατε κάποιε εξηγήσει για να δείτε τι κάνει ο εισηγητή, ο σχεδόν εισηγητή, ο συντονιστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ πρέπει να σα πω ότι είναι μένα εδώ, είναι η πρώτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009, εκπροσωπώ του πράσινου, αλλά Άρχισα στην αρχή της θητείας μου με τον ε, φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη στην ε, ε, ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Και για λόγους εθνικής, εσωτερικής πολιτικής στην Πορτογαλία άλλαξα. Αλλά είμαστε μαζί στην ίδια επιτροπή. Εγώ πάρα πολύ καλά όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ καλά σε δύο μας που συνεργαζόμαστε πολύ σωστά. Όπως και ο Αντώνιο που πρέπει να πω ότι ήταν ο ισχυρό συγητής της εισήγησης στην οποία σας παρουσιάσω, καθώς και άλλοι συνάδελφοι εδώ παρόντες με τους οποίους υπάρχουν στις διάφορες επιτροπές. Οι πλειοψηφίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου πολλές φορές πρέπει να πω ότι πολλές φορές είναι ανεξάρτητες και ανέλπιστες σύμφωνα με τις στατιστικές. Πρόκειται για μεταβλητή γεωμετρία η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εδώ εκπροσωπείται πολύ παλά και πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει στο Κοινοβούλιο πλειοψηφία κέντρο δεξιάς η Επιτροπή, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ οι φιλελεύθεροι όπως και η κυρία ε, Βίξτρομ ψηφίζουν πιο προοδευτικά όπως και η αριστερά. Και αυτό γίνεται για τις περισσότερες εκθέσεις που συζητούν Και Κυρίως εγώ για τη δική μου εισήγηση που αφορά την μετεγκατάσταση και μετακίνηση των προσφύγων, πρόκειται για δύο εκθέσεις τελικά, είχα την τύχη να έχω μια πλειοψηφία που υποστηρίχθηκε από τους ε, ε, κομμουνιστές, τους Έλληνες και τους Κυπρίους μέχρι τους συντηρητικούς, τους Βρετανούς που εκπροσωπεί εδώ ο συνάδελφος Τίμωθη Κίρχοπ. Τώρα, πώς συνέβη κάτι τέτοιο. Και τώρα θα συνεχίσω αγγλικά, διότι θα προσπαθήσω σε δύο λεπτά να σας εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε με την κατάσταση και μετακίνηση προσφύγων και τι προσπαθούμε να κάνουμε μέσα τη εισήγηση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ίσως δεν είναι εύκολο να καταλάβετε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας εξηγήσω. Λοιπόν, Γνωρίζετε ότι υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες, ετούντες άσυλο, που μπορεί να είναι πρόσφυγες μέσω του καθεστώτος προσφύγα που καθορίζει η Πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες ή ε, και πρόσφυγες με την ευρία έννοια διότι ξεφεύγουν από ένα πόλεμο ή διώκονται και μετά έχουμε πρόσφυγες με την πιο αυστηρή τους έννοια, άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν καθοριστεί ως τέτοια από την ύπατη αρμοστία ε, βάσει της ε, σύμβασης της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι κάποιος ο οποίος ε, έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου δεν μπορεί να θεωρείται πρόσφυγα και δεν ε, τη, χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα βάσει της σύμβασης. Εντός λοιπόν της ομάδας των προσφύγων υπάρχουν διάφορες υποομάδες. Ανάλογα με τις τρεις λύσεις που ε, μπορεί να ε, δοθούν σε κάποιον ο οποίος θεωρείται πρόσφυγας. Μπορεί να επιστραφεί στη χώρα του, που είναι το, η περίπτωση των 90% των προσφύγων. Αυτό θέλουν να κάνουν ούτως ή άλλως. Δεν φεύγουν με τη θέλησή τους από τη χώρα. Ε, μπορεί να φεύγουν διότι διώκονται. Το 90% θέλει να επιστρέψει λοιπόν στη χώρα του και σε πολλές περιπτώσεις όταν ε, η σύραξη για παράδειγμα υποχωρεί επιστρέφουν. Αυτό υποθέτουμε ότι θα γίνει και με τους σύρους πρόσφυγες ε, όταν σταματήσει η ένοπλη σύραξη και ελπίζουμε ότι θα γίνει σύντομα και θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Επίσης, οι πρόσφυγες μπορούν να μείνουν στη χώρα στην οποία έχουν πάει, που είναι συνήθως μια γειτονική χώρα, όπου συνήθως βρίσκουν την ίδια εθνοτική ομάδα, την ίδια θρησκευτική ομάδα ή και την ίδια γλωσσική ομάδα ε, τη, με, που, με τη χώρα από την οποία προέρχονται. Ε, αυτό είδαμε και για παράδειγμα στη Συρία πριν από τον πόλεμο στη Συρία υπήρχαν πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονταν από το Ιράκ ή και Παλαιστίνοι οι οποίοι είχαν ζήσει στο Ιράκ και με τον πόλεμο στο Ιράκ μεταφέρθηκαν στη Συρία. Και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στη Συρία, διότι η Συρία δεν ε, έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να εργαστούν εκεί, δεν μπορούσαν να ε, έχουν μόνιμο καθεστώ πρόσφυγα και σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να έχουν και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ε, ή σε σχολεία. Κάποιοι που είχαν κάποια χρήματα, γιατί προέρχονται από τη Βαγδάτη ή από άλλες πόλεις, ε, εξόδευαν τα χρήματά τους και μετά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στις κοινότητε προσφύγων, τα οποία είδαμε και η διεισόμαση στην περιοχή της Τζαραμάνη στη Δαμασκό ή και στα βόρεια της Συρίας, στην ε, περιοχή του Αλχάζακε, όπου εκεί υπήρχαν πρόσφυγες χωρίς χρήματα και έκαναν μικροκλοπές, ε, πορνεία, παιδική εργασία και ούτω καθεξής. Για μία άλλη υποδομάδα προσφύγων δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ε, πρέπει να τους δοθεί δικαίωμα σε νέα ζωή σε μια άλλη χώρα. Αυτό καλείται με την κατάσταση. Και περίπου 200.000 πρόσφυγες ετησίως χρειάζονται με την κατάσταση. Επομένω, έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγε παγκοσμίω και αναφερόμαστε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ε, προσφύγων. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σκοτωθούν, ε, θα του σκοτώσουν αν επιστρέψουν στη χώρα του και δεν μπορούν να μείνουν και στη χώρα που βρίσκονται, διότι η χώρα δεν έχει προσυπογράψει τη σύμβαση τη Γενέβη και υπάρχει και πρόβλημα στο στρατόπεδα προσφύγων. Ε, έχουμε βιασμού, μπορεί να συμβεί παρά το γεγονό ότι υποτίθεται ότι προσπαθούμε να του έχουμε στο δυνατόν πιο ασφαλεί. Ορισμένες φορές ζουν και σε χώρους που είναι ε, κίνδυνοι. Υπάρχουν πλημμύρες, ε, πυρκαγιές και κάποιοι ε, πάσχουν από πολύ κοινέ ασθένειες, ε, ε, διαβήτη για παράδειγμα και πρέπει να ε, τύχουν νοσηλεία σε άλλη χώρα. Τι κάναμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετοιμάσαμε δύο διαφορετικές εκθέσεις. Μία έκθεση με διαδικασία συναπόφασης, που σημαίνει ότι θα είναι πρόταση νομοθεσίας και θα ενταχθεί στην νομοθεσία και αυτό αφορούσε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων που ε, βοηθά ε, τα κράτη-μέλη για να στηρίξουν τους πρόσφυγες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε μετεγκατάσταση περίπου 5.000 προσφύγων. Σκεφτείτε ότι έχουμε 200.000 ε, ε, παγκοσμίως και εμείς βοηθούμε μόνο 5.000. Ποιος δίνει περισσότερους, οι Ηνωμένε Πολιτείε, 80.000. Μετά έχουμε Καναδά, Αυστραλία, Βραζιλία, Χιλή και άλλες χώρες. Επομένως, 100.000 πρόσφυγες από τους 200.000 που πρέπει να μετεγκατασταθούν κάθε χρόνο ε, μετεγκαθίστανται. Αυτό σημαίνει το ότι το 50% του προβλήματος το έχουμε λύσει. Και αν η Ευρώπη έκανε όσα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, θα ήταν λυμένο το πρόβλημα. λιμένο πρόβλημα στον κόσμο της μετανάστευσης και του ασύλου είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επομένω ε, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Η Βρασιλία και η Χιλή βέβαια αυξάνουν συνέχεια τον αριθμό των προσφύγων και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει όμως ε, ε, στο νέο κανονισμό και κάποια μέτρα για να βοηθήσουν αυτούς που δεν έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα. Οι 17 χώρες είχαν πρόβλημα με τη μετεγκατάσταση. Ε, στο μεταξύ, για παράδειγμα, η Ισπανία ξεκίνησε μετεγκατάσταση ε, και αν προέρχεστε από μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει πρόγραμμα μετεγκατάσταση, θα πρέπει να ρωτήσετε τον Υπουργό Ιστορικών Υποθέσεων γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα μετεγκατάσταση. Και αν απαντήσουν ότι αυτό έχει να κάνει με οικονομικού μετανάστε και ετήντου άσυλο, θα πρέπει να του εξηγήσετε ότι δεν έχει καμία σχέση, πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Και μετά είχαμε μια άλλη έκθεση που είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και είχε άλλα θέματα. Και θα πρέπει να, να, να σας τα εξηγήσω λίγο για να καταλάβετε τη διαδικασία. Εγώ ήρθα ε, το 2009 εδώ, 9, ως Ευρωβουλευτής που δεν έχει καμία σχέση με τις εκθέσεις. Και τελειώνει η έκθεση και ως αδαής θεώρησα ότι τελείωσε ε, η δουλειά μου. Όχι, τότε ξεκινάει η δουλειά, γιατί η έκθεση στο Κοινοβούλιο είναι μισή δουλειά. Μετά η έκθεση πάει στο Συμβούλιο και μετά ξεκινάμε την άλλη μισή δουλειά. Στο Συμβούλιο έχουμε εκπροσώπους των κυβερνήσεων, άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα της μεταγκατάστασης ή κάποιοι που δεν γνωρίζουν καθόλου την μεταγκατάσταση και περιμένουν οδηγίες από την πρωτεύουσά τους που μπορεί οι υπουργοί τους να γνωρίζουν ή να μην γνωρίζουν τι γίνεται με τη μεταγκατάσταση. Περάσαμε τέσσερις προεδρίες, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία και Ουγγαρία. Και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία δεν υπήρχε σχεδόν καμία Πρόοδο για το θέμα αυτό και δεν έγινε γιατί ο, δεν βοήθησε ο Μασί Πιντάλγο γιατί προσπάθησε πάρα πολύ να βοηθήσει στη διάρκεια τη ισπανική προεδρία και τα κατάφερε. Εν τέλει, ανέλαβε τα ημία η Ιδανική Προεδρία και τα κατάφερε. Και η ηρωνία, και αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα, ε, είναι ότι οι Δανείοι είχαν δικαίωμα να μην συμμετέχουν στην πολιτική αυτή, είχαν opt-out και όλες οι άλλες χώρες θα λάβουν οικονομική στήριξη για αυτές τις πολιτικές οι Δανείοι δεν θα λάβουν ούτε έλαμβαναν ούτε σεντ ούτε ευρώ στήριξη από αυτό το πρόγραμμα. Και παρόλα αυτά ήταν αυτοί που κατάφεραν να τελειώσουν το, ε, το θέμα επειδή η Προεδρία είναι αυτή που έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει το θεματολόγιο του Συμβολίου. Και γιατί αυτό, γιατί τότε ήρθε κάποιο από την Κοπεχάγη που ήξερε τι συμβαίνει με του πρόσφυγε. Ήξερε ότι με την κατάσταση των προσφύγων είναι μια μακροβόρα διαδικασία οι πρόσφυγες έχουν προβλήματα με τη γλώσσα. Ε, μπορεί να είναι μια ε, επώδυνη διαδικασία η μεταφορά τους. Επομένως, μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα με τους πρόσφυγες από ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, γιατί είναι πιο άτακτη η μετανάστευση αυτή. Αν και πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικώς είμαι υπέρ της μετανάστευσης ως πολιτικός, είμαι ε, πάγια θέση μου είναι υπέρ της μετανάστευσης ε, και για τους οικονομικούς μετανάστες. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει μεγάλο φάσμα θέσεων, αλλά πρέπει να σας πω ότι για τους πρόσφυγες κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και μετά που εγκρίθηκε η έκθεση, με πολλούς συναδέλφους, σχεδόν γκρινιάζαμε μπορώ να σας πω, συνέχεια στο Συμβούλιο, αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, τους γκρινιάζαμε, τους πιέζαμε κάθε δυο μένα προσφορικές ερωτήσεις, ε, και ο Τίμωθη Κύρκοφ, παρά το γεγονό ότι έχουμε τελείω διαφορετικέ θέσει, είπε κάποια στιγμή στο Συμβούλιο ότι δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει ο Ταβάρε, αλλά κάντε το, επιτέλου, τελειώστε το. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε και με αυτό θα ολοκληρώσω ότι η συναπόφαση στις συνθήκες σημαίνει ε, ότι επειδή δεν υπάρχει και καταληκτική προθεσμία για τη συναπόφαση, ότι το Συμβούλιο μπορεί να εφαρμόσει αυτό που λέμε εμείς στην ε, ε Πορτογαλία, δικαίωμα της ε, ανησυχηρίας του συρταριού. Τι κάνουμε, παίρνουμε την νομοθεσία, τη βάζουμε στο συρτάρι και δεν κάνουμε τίποτα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι βέτο αυτό. Και αυτό λέω, λέω ότι ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία, η οποία ορισμένε φορέ κολλάει, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι σκανδαλώδο και καλό είναι να το παρακολουθούν και οι δημοσιογράφοι και κάποια στιγμή να ενημερώσουν του πολίτε, γιατί καθυστερεί η νομοθεσία ε, στα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βέβαια αυτή είναι η συζήτηση μιας άλλης ημέρα. Ευχαριστώ κύριε Ταβάρης. Ναι, αυτή είναι μια νέα ολόκληρη συζήτηση για τη μεθοδολογία. Ο κύριος Τίμωθη Κίρκοπ μάλλον γνωρίζει πολύ καλά τη μεθοδολογία, διότι ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κίρκοφ είναι συντονιστής. Μέχρι τώρα ακούσαμε εισηγητέ. Εσείς ο συντονιστής λοιπόν, πώς βλέπετε το θέμα αυτό και, και για το μέλλον από πλευράς της δικής σας πολιτικής ομάδος ε, αλλά και, τη, και προσωπικός. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Οι παρατηρήσεις μου νομίζω ότι θα είναι ένα ευρύτερο όραμα. Δεν θα σας δώσω απλώς ε, συγκεκριμένα στοιχεία για νομοθεσία ή προτάσεις νομοθεσίας. Κάτι θυμάμαι ότι είχα πει. Μάλλον τους είπα ότι τελειώνετε με τον Ταβάρες. Δεν σας είπα τελειώνετε το ζήτημα, αλλά τέλος πάντων. Πέρα από τα αστεία, ε, πράγματι συνεργαζόμαστε, νομίζω σχετικά καλά και για πολλά πράγματα, παρά το γεγονό ότι πολιτικώ έχουμε διαφορετικέ ιδεολογίε και αυτά είναι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχει μια συνενετική διάθεση σε ευαίσθητα ζητήματα όπω αυτά. Και πολύ συχνά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι το οποίο θα ήθελα να πω, ε, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξή. Ε, νομίζω ότι δεν μιλάμε αρκετά για τη μετανάστευση. Νομίζω ότι δεν μιλάμε ξεκάθαρα για τα θέματα αυτά, ε, τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε. Διότι αν θέλουμε να αποφύγουμε και την κακή πλευρά της αντίδρασης των ανθρώπων απέναντι στο άσυλο, ε, ε, μία λύση θα είναι να το συζητήσουμε. Οι πολιτικοί οι οποίοι εκλέγονται με δημοκρατικό τρόπο και ελπίζω ότι έχουν ισορροπημένη και ευαίσθητη προσέγγιση θα πρέπει να μιλούν περισσότερο και όχι λιγότερο για τα θέματα αυτά. Το, το άσυλο με ενδιαφέρει εδώ και αρκετά χρόνια και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις της κυρίας Βίξτρομ διότι και εγώ ήμουν υπεύθυνο ε, για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα προσφύγων της Βοσνίας ε, των Ηνωμένων Εθνών στη δεκαετία του 90 και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές χώρες συμμετείχαν και ήταν καταμερισμένη η ευθύνη για το θέμα αυτό και τη θεώρησα και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είναι μια πρωτοβουλία που ε, θα μπορούσε να συνεχιστεί και τώρα όταν ασχολούμαστε με διάφορες δύσκολες περιοχές του κόσμου. Αλλάζει το τοπίο παγκοσμίων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μου τα ε, ε, μοντέλα της μετανάστευσης έχουν αλλάξει ε, πολύ από, ακόμα και από τη δεκαετία του 90. Ο κόσμος ταξιδεύει πιο μακριά, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερους αριθμούς και αυτό φυσικά αποτελεί πρόκληση για τους πολιτικούς και φυσικά οι, χώροι, οι χώρες που έχουν προβλήματα, οι περιοχές που έχουν προβλήματα είναι πολύ περισσότερες πλέον. Ε, με την άφηξη δε της τρομοκρατίας, των ε, οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων που είναι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι ποτέ, ε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε υπαλλήλου που ασχολούνται με τη μετανάστευση και με πολιτικού που ασχολούνται με τη μετανάστευση και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία στον τομέα αυτό. Όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο Εστερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσπάθησα να εφαρμόσω πολιτικέ ε, στον τομέα τη μετανάστευση, τι οποίε θεωρώ αυστηρέ αλλά δίκαιε και θα πρέπει να ε, εξετάζονται τα όλα με διαφάνεια. Και στη χώρα μου αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε. Πάντα θεωρώ ότι ο Υπουργό που ασχολείται με θέματα μετανάστευση και ασύλου δεν θα πρέπει να έχει μόνο διπλωματία, αλλά θα πρέπει να επιδεικνύει και ανθρωπιά. Και είναι πολύ σημαντικό ε, να δείξουμε ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες ή με τα κριτήρια, όπως για παράδειγμα τη σύμβαση του 51 για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι οι νεοαφιχθέντες, αλλά οποιοδήποτε καταχράτε τους κανόνες και εκμεταλλεύεται ανθρώπους θα πρέπει να τιμωρείται. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θέλουμε να τα βλέπουν με θετικό πνεύμα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να τα συζητούν καν αυτά τα ζητήματα και λένε ότι οι πολιτικοί που τα συζητάνε είναι ρατσιστές ή ακραίοι αλλά νομίζω ότι το να χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς ε, δεν ε, ε, ευνοεί κανέναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το άσυλο, είναι σημαντικό θέμα των καιρών μας και θα πρέπει να έχουν οι πολίτες τον τελικό λόγο. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι οι πολιτικοί... προσμετρούνται από τις αποτυχίες τους και τις επιτυχίες μας και ασχολούμαστε με αυτό και ελευθερεύει ο κίνδυνος να χάσουμε στη συζήτηση αυτή από ακραία στοιχεία. Και αυτό το οποίο προσάπτω στους Ευρωπαίους πολιτικούς είναι ότι δεν το συζητούν αρκετά. Στη μελλοντική μας νομοθεσία λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε τι αποτελέσματα θέλουμε να έχουμε. Μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε εδώ τις ευαισθησίες μας και τα προβλήματά μας, αλλά θα πρέπει να τα δούμε λίγο πρακτικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, στεναρό συνεκτικό σύστημα και να πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι χώρες όπως η Μάλτα και η Ελλάδα που δίνουν ε, μάχη για αυτά τα ζητήματα θα ε, βοηθηθούν από τους υπολείπους το να έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία και λιγότερη ευελιξία σίγουρα δεν θα μας βοηθήσει. Επίσης, εγώ ήμουν ε, και υπουργό για ε, ρατσιστικές ε, υποθέσεις και θέματα φύλου και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για τις σχέσεις με τις διάφορες φυλές που έχουμε στις χώρες στις οποίες έχουμε πρόσφυγες ε, γινόμαστε λίγο πιο ανεκτικοί με την ανοιχτή οικονομία, αλλά θα μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα μόνο αν είναι ρεαλιστικοί και βιώσιμη. Ε, οι πρόσφυγες αναζητούν βέβαια μια καλύτερη ζωή, αλλά η μετανάστευση δεν είναι δικαίωμα για όλους απαραίτητα και αυτοί που ε, πλήττονται περισσότερο από την παράνομη μετανάστευση είναι οι ίδιοι παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται με τις φρούδες ελπίδες μιας ε, καλύτερης ζωής χωρίς να έχουν καμία εγγύηση ότι θα ζήσουν με καλύτερο τρόπο και θα έχουν θέση εργασίας και βλέπονται, τους βλέπουμε πολύ αρνητικό μάτι η υπόλοιπη κοινωνία και Όλη αυτή η ψευδής αλληλεγγύη υποσκάπτει αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και τα κράτη-μέλη κάνουν πάρα πολλά πράγματα στο όνομα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας και ουσιαστικά όλα αυτά είναι εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Οι προκλήσεις του Ευρωπαϊκού ε, Συστήματος Ασύλου ε, αφορούν ε, θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακόμα και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυσκολευόμαστε να συμβάσουμε τι απόψει των 7 πολιτικών μα ομάδων. Πότε, πότε τα καταφέρνουμε, όπω είπαμε. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι να προσπαθούν 27 να συμφωνήσουν ναι, για αυτά τα θέματα. Και 27 χώρε μέλη έχουν και διαφορετικέ κοινωνικέ, γεωγραφικέ, περιφερειακέ, οικονομικέ ε, πραγματικότητε και αυτό το οποίο συζητούμε εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπόφευκτα είναι διαφορετικό από αυτό που θα συζητήσει η Ισπανία ή η Ολλανδία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά τη μετανάστευση, ούτε είμαστε κατά της ε, ένταξη και τη αλληλεγγύη. αλλά... Ε, το κάθε διαφορετικό σύστημα σημαίνει ότι κανένας ε, δεν αντιμετωπίζει το θέμα στη χώρα του με τον καλύτερο τρόπο. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις βασικές θεμελιώδεις αρχές και θα πρέπει να νομοθετούμε με τρόπο ο οποίος θα είναι εύκολος ε, στην εφαρμογή του και απλός. Ε, λέμε ότι θέλουμε μια νέα προσέγγιση για την ε, μετανάστευση, αλλά εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει κυρίως να ασχοληθεί με το να διαπιστώσει κατά πόσον οι ευρωπαϊκές χώρες ε, μεταχειρίζονται με δίκαιο τρόπο τους ε, ετούντες άσυλο. Στη Σύμβαση ε, για τους πρόσφυγες και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπάρχουν τα πάντα και το να δημιουργήσουμε νέους κανόνες νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί με την ουσία. Οι κυβερνήσει πρέπει να τηρήσουν τι δεσμεύσει του και να μεταχειρίζονται του ανθρώπου με αξιοπρέπεια. Και νομίζω ότι εδώ και καιρό έχουμε χάσει το στόχο μα και προσπαθούμε συνεχώ εδώ να δούμε πόσε ώρε, ε, πόσα έγγραφα θα πρέπει να διεκπεραιώνονται και ποιο θα πρέπει να είναι αρμόδιο γιατί. Τσακωνόμαστε για όλα αυτά και σε κάποια κράτη-μέλη φοβόμαι ότι ο τίντε άσυλο που αναζητούν μια καλύτερη ζωή δεν έχουν πού να κοιμηθούν, πού την κεφαλή κλείνε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το θεωρούμε επωνίδιστο στον 21ο αιώνα. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ως συντονιστής της ΓΚΟΕ, τη Ανατολική Αριστερά, έχετε το λόγο. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση όσον αφορά αυτό το τόσο πολύπλοκο θέμα. Και τους ε, πάρα πολύ πολύπλοκους τρόπους για να καταλήξουμε σε ένα τέλος. Ευχαριστώ. Εγώ κύριε Πρόεδρε άρχισα ως καθηγητής και όταν βλέπω μια τάξη τόσο ήσυχη Σκεφτόμουν παλιότερα από ένα αστείο για να ξυπνήσω τους μαθητές. Εν δεν ξέρω αστεία, αλλά παρακαλώ, ακούστε με, ε, κάντε λίγη υπομονή, μην κοιμηθείτε. Θα ξυπνήσουμε. Θα ξυπνήσουμε μετά ούτως ή άλλως μετά από τις ερωτήσεις που θα τεθούν μετά από τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων. Φαίνεται λοιπόν ότι όλοι όσοι πήραν το λόγο στο πάνελ εξήγησαν για ποιους λόγους επέλεξαν να ασχοληθούν με το θέμα το οποίο συζητείτε εδώ από σήμερα το πρωί. Ποιος είναι ο δικός μου λόγος. Εγώ είμαι Κύπριος, ένα μικρό νησί στην ε, Ανατολική Μεσόγειο, με όχι πολύ πληθυσμό, αλλά που έχει μεγάλη ιστορία στα θέματα χωρίς ασύλου. Πρώτα απ' όλα, διότι και το ίδιο το νησί μας, όπως ξέρετε, ήταν ε, θύμα επειδή το 1974 και εισβολής, μετά την οποία ε, μετατοπίστηκε το 1 τρίτο του πληθυσμού και το, αυτό το τρίτο ζύος πρόσφυγε σήμερα. Δεύτερον, εξαιτία γεωγραφικής θέση του νησιού μας. Από τότε προσχώρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 η Κύπρος είναι η πύλη, αν θέλετε, για πολλούς ε, ε, μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Και όπως και η Μάλτα και η, Ευρώπη, και η, Μάλτα και η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες, η Κύπρος είναι μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες εισέρχονται μετανάστες και πρόσφυγες για να προχωρήσουν περαιτέρω στα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ κυρίως ασχολούμαι με το θέμα της ε, αλληλεγγύης στον τομέα της χορήγης ασύλου. Η αλληλεγγύη είναι ένας όρος που ακούγεται ωραία, που όλοι θέλουμε να τον ακούμε. Αλλά είναι μάλλον ε, σλόγγαν εάν δεν του δώσουμε κάποιο περιεχόμενο και δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Όπως ακούσατε και από άλλους συναδέλφους, εξαιτίας των χαρακτηριστικών του, το σύστημα του του Δουβλίνου δεν προβλέπει ένα ε, δίκαιο σύστημα για τους ετούντες άσυλο. Δίδεται ευθύνη για την εξέταση των ετοιμάτων που υποβάλλονται στην πρώτη χώρα εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη χώρα εισδοχή, σαν την Κύπρο, σαν τη Μάλτα, σαν την Ελλάδα. Και έτσι ε, υπάρχουν δυσανάλογα αιτήματα από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως υπάρχουν και τρομερά προβλήματα ένταξης και ενοποίησης. Ε, Εξορισμού λοιπόν δεν είναι δίκαιο το σύστημα αυτό και είναι τέτοια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν ένα παρεμφερές σύστημα ασύλου. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι δεν παρέχεται υψηλό σύστημα προασίας ε, από σε πολλές χώρες. Θα ήθελα λοιπόν ε, το 2014 να πω ότι θα κάνει η Επιτροπή ένα check-up στο όλο σύστημα αυτό για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Στο μεταξύ διάστημα παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερο σημαντικό να μιλήσουμε για αλληλεγγύη όχι μόνο σαν έναν όρο αλλά σε ένα, μια αρχή που πρέπει να τεθεί στην πράξη σε εφαρμογή και πραγματικά να εφαρμοστεί. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση για να έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό, δεν έχουμε ισχυρό σύστημα διεθνούς προστασίας, δικαιωμάτων και ελευθεριών εάν τους αδύναμους κρίκους της αλυσίδας που έχουμε τους παραγνωρίζουμε. Είναι υποχρέωσή μας να βρούμε τους σωστούς τρόπους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την αλληλεγγύη, δεδομένου ότι θα πρέπει εντός του συστήματος του Δουβλίνου να βρούμε τρόπους για να αμβλύνουμε όλες τις δυσάρεστες πλευρές του κανονισμού του Δουβλίνου. Στον τομέα του ασύλου, ήθελα να υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε η σχετική έκθεση ώστε να μπορέσουν να έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και τους κανόνες που θα υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη που έχουν δυσανάλογα αιτήματα χορήγηση ασύλου. Μόνο εάν βελτιώσουμε τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών θα εξασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίζονται και θα προστεύονται πλέον τα δικαιώματα των ετούντων ασύλου. Θα ήθελα τώρα, Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για το τι θέλουμε να δώσουμε ως περιεχόμενο στην ε, αλληλεγγύη. Υπάρχει το γραφείο Ιάσο, το οποίο νομίζω ότι παίζει θεμελιώδη σημασία ρόλο στον ε, προσπάθεια που καταβάλουμε. Είδαμε ότι ενήργησε το Ιάσο στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο και το ΕΑΣΟ. Το κέντρο αυτό είναι πολύ σημαντικός φορέας στον τομέα αυτό και δίνει μεγάλη υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Από αρχική ε, εντόπιση των προβλημάτων που υπάρχουν, την, ετοιμότητα για τη διαχείριση κρίσεων, την έγκαιρη προειδοποίηση, τον συντονισμό, την πρακτική χορήγηση βοήθειας, την κατάρταση, τη διαχείριση ε, προγραμμάτων ε, και βοήθηση με ειδικέ ομάδες προετοιμασίες και υποστήριξη στην προετοιμασία των ε, και στην σωστέ σχέσει που πρέπει να υπάρχουν με την χώρα καταγωγή των ετούντων άσυλων. Ε, θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με τις διεθνείς οργανώσεις επίσης και με την κοινωνία των πολιτών για να είναι η συνεργασία αποδοτική, να ανταλλάσσονται ε, γνώσεις και εμπειρίες και για να βοηθηθούν οι χώρες οι οποίες υφίστανται μεγάλες και δυσανάλογες πιέσεις. Ο Ρούι ανέφερε προηγουμένως διάφορα κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούμε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε με όλα αυτά τα προγράμματα. Ένα άλλο στοιχείο της ελληνικής είναι τα διάφορα κοινοτικά κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το, να υλοποιηθούν οι στόχοι του ασύλου. Στα πλαίσια των ε, αυτή τη πολιτική θα πρέπει να έχουν σωστή ενημέρωση οι διάφορες κυβερνήσεις, να ξέρουν ποια είναι η κοινοτική χρηματοδότηση, ώστε να επικουρώνται οι χώρες οι οποίες έχουν ένα πρόγραμμα υποστήριξης και αυτό τι σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε λιγότερα προγράμματα, αλλά με τη σωστή χρηματοδότηση, ώστε να έχουμε θετικές επιπτώσεις. Τα δύο τελευταία στοιχεία τα οποία ήθελα να σας αναφέρω, δίδοντάς σας πρακτικά παραδείγματα αλληλεγγύης, είναι πρώτα απ' όλα η χρησιμοποίηση μίας ε, κοινή διαδικασίας για τη χορήγηση ασύλου και το θέμα της μετακατάστασης και της ε, αποκατάστασης η μετεγκατάσταση, το relocation, είναι αν θέλετε η αδελφή έννοια με το resettlement που ανέφερε ο Ρούι Ταβάρες. Το πρώτο θέμα είναι θέμα εφαρμογής της πολιτικής αλληλεγγύης που έχουμε εάν έχουμε η μεγάλο αριθμό ε, ε, ασύλου η κοινή διαχείριση και επεξεργασία όλων αυτών των ετοιμάτων και η προετοιμασία των πρώτων σταδίων συνέντευξης και ε, διοικητικών ε, διαδικασικών είναι κάτι το οποίο μειώνει το άχθος και το οικονομικό κόστος, μειώνει το χρόνο ε, ανταπόκρισης στα αιτήματα των προσφύγων και εξασφαλίζει τα δικαιώματα και την προστασία τους. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν ε, να ληφθούν οι σωστέ αποφάσει το μέσο αυτό που προβλέπεται να μπορέσει να θέσει εφαρμογή σύστημα. Δεύτερον, το θέμα του relocation, τη επανεγκατάσταση. Επίση και τη μετακίνηση είναι κάτι το οποίο ε, έχει γίνει βάση ενό πιλωτικού σχεδίου στη Μάλτα που λέγεται Γιουρίμα και μπορεί να αποδείξει πόσο εύκολα μπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη και να δώσει κατάλληλους όρους για τους πρόσφυγες. Η Επιτροπή ε, έχει την πρόθεση να προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό relocation ώστε να επικουρούνται οι χώρες οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε, ακόμη δεν υπάρχει σχετική και συγκεκριμένη πρόταση, διότι κάποιε χώρε έχουν επιφυλάξει ότι πιστεύουν ότι κάποιοι θα το χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό για να μεταφέρουν σε κάποιον άλλο τις του και να μην τι επομιστούν. Πρόκειται όμω για ένα μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσει όπου είναι δυσανάλογα μεγάλο ο αριθμό των ετούντων άσυλο σε σχέση με τι δυνατότητε που έχει ένα κράτο μέλο να υποδεχθεί πρόσφυγες. Η relocation είναι ε, πρέπει να είναι επωφελής και για το κράτος υποδοχής και για τους ετούντες άσυλο από τη στιγμή που αξιολογεί σωστά κάποια θέματα σημαντικά όπως το ΑΕΠ, τον πληθυσμό, τις δυνατότητες απορρόφησης της χώρας υποδοχής και τις δυνατότητες συνεργασίες. Ως επίλογο θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταδείξουμε την αλληλεγγύη μας και από απλά λόγια να την κάνουμε έργα. Το, μές το αυτό το οποίο λείπει δεν είναι λόγια, είναι η πολιτική βούληση. Φαίνεται ότι είναι για κάποια κράτη-μέρη κάποια ε, θέματα να τα κατανοήσουν σωστά κάποιες χώρες μέλη και μπλοκάρουν την κατάσταση στο Συμβούλιο και πρέπει να πω ότι σήμερα με μεγάλη χαρά συμμετέχω στο δικό σας σεμινάριο και αναμένω με ενδιαφέρον τις ερωτήσεις που θα μου υποβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ. Thank so Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Και η Ιταλία είναι χώρα ασύλου και προσφύγων. Εξ ονόματος λοιπόν των ε, συντονιστών, ως συντονιστής ε, της Ομάδας Ελευθερίας και Δημοκρατίας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με τις ε, θετικές αξιολογήσεις για τα όσα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και ένας Θεός ξέρει πόσο ανάγκη το είχαμε. Εμείς ως ευρωσκεπτικιστές θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου δεν θα ήθελα τώρα να είμαι πολύ επικριτικός και σκληρός και να πω ότι ήταν απόλυτη αποτυχία, αλλά δεν απέχουμε και πολύ. Και η δήλωση αυτή ε, επιβεβαιώνεται και από τις ειδήσει που μας στάνουν ακόμα και σήμερα από τη Σουηδία. Αλήθεια δεν είναι ότι η Σουηδία ζητά να ανακληθούν όλες οι θεωρήσεις εισόδου για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Βόσνια, Κωσυφοπέδιο, Αλβανία ε, και ούτω καθεξής όλες, όλες αυτές οι φωνές του ενθουσιασμού και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και μια χώρα υποδοχής, μια πολιτισμένη χώρα ε, και σίγουρα φιλελεύθερη όπως είναι η Σουηδία, ζητά να ανακληθούν οι άδειε, διότι βρέθηκε, βρέθηκε ενώπιον ε, μια δυσκολίας... ενός πραγματικού φαινομένου που πρέπει πρώτος να το ε, αντιμετωπίσει. Έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμό των πλαστών αιτήσεων ασύλου, ψευδών αιτήσεων ασύλου. Και είναι κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε τόση ώρα. Ε, το γνωρίζουν βέβαια οι συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι είναι το εγνωσμένου κύρους και σίγουρα τα γνωρίζουν αυτά, αλλά το θέμα είναι αν οι δέσμοι μέτρων για το άσυλο που θα ψηφίσουμε και θα ε, συζητήσουμε αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αυτόν τον κίνδυνο. Και θα ήθελα ε, να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί ακούσαμε όλες τις απόψεις και που στο θέμα αυτό διέπονται και από ένα φιλοσοφικό, θεολογικό πνεύμα. Ένας μεγάλος κοινωνιολόγος, ο κ. Παρέτο, θα είχε πει ότι είναι αλτρουισμός. Εγώ ε, δεν είμαι τόσο ε, υψηλών φρονημάτων, με κάθε σεβασμό για όσους θεωρούν ε, ε, τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από μένα, είναι λίγο υποκριτική η στάση μας. Η πραγματικότητα μας επιτάσσει τρεις ερωτήσεις και οι ερωτήσεις μου είναι εξή. Καταρχάς, πώς μπορούμε να δηλώνουμε ότι αυτός ο ευγενή θεσμό, διότι ο θεσμός του ασύλου δεν έχει ξεκινήσει από τη Γαλλική Επανάσταση. Είναι θεύμα πολιτισμού, αν, έρχεται απαρχαιότητά των χρόνων. Εφαρμόστηκε στην πράξη τα προβλήματα επέτρεψαν για παράδειγμα στις οργανώσεις του εγκλήματος που κάνουν ε, παγκοσμίω διακίνηση ναρκωτικών να χρησιμοποιήσουν το άσυλο για να κάνουν τις δουλειές τους. διότι όταν ε, οι ταλέποροι πρόσφυγες ε, έφευγαν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και έμπαιναν στις βάρκες για να φτάσουν στις Ιταλικές ακτές, τους υποδέχονταν μέσα στη μέση της νύχτας από τη μέλη της Δράγκετα ή έφταναν στις αυτές της Σικελίας και τους υποδεχόταν η μαφία και τους έδιναν και τη διεύθυνση για το που πρέπει να αποτανθούν. Και εκεί τους στρατολογούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν μικροδιακίνηση ναρκωτικών, διότι αυτές οι οργανώσεις δεν κάνουν πλέον διακίνηση απευθείας, την ε, δίνουν σε, ε, σε αυτούς τους ε, ταλέπορους που έρχονται από όλες τις γωνιές της γης. Πρόκειται λοιπόν για όλη αυτή τη συζήτηση, συζητάμε όλη αυτή την ηθική και νομική ε, ε, διαδικασία, τον ορισμό των προσφύγων. Ε, στην πραγματικότητα είναι όλοι αυτοί οι καημένοι, τα λέποροι που έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να επιβιάσουν. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη ηθική επιταγή διότι αν συγκρίνουμε τον αριθμό ε, όντως των ανθρώπων που ζητούν άσυλο για οικονομικούς λόγους ε, με τον, αριθμό, τον μικρό αριθμό των ανθρώπων που διώκονται, θα πρέπει λοιπόν να μην αφήνουμε να τους εκμεταλλεύονται. Στο πακέτο λοιπόν υπάρχει μια διάταξη την οποία θεωρώ θετική και αυτό είναι η διαδικασία της Eurodac. Επιτέλους, αν και κατόπιν εορτής, επιτρέπεται στις αστυνομικές δυνάμεις ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδεθούν σε μια βάση δεδομένων και να λάβουν σε πραγματικό χρόνο διακριτικά αποτυπώματα. Αυτά μέχρι τώρα δεν συνέβαινε. Ο καθένας αναγκαζόταν να διαχειριστεί την κατάσταση μόνος του. Πλέον μπορεί η αστυνομία ε, που θέλει να εντοπίσει έναν ε, παράνομο μετανάστη ε, να δει αν ε, δρά ε, παράνομα σε άλλες περιοχές ή αν κάποιος που κάνει αίτηση ασύλου έχει κάνει αίτηση και σε άλλες χώρες. Ξέρετε τι προβλήματα υπάρχουν όταν υπάρχουν πολλές αιτήσει σε διάφορες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα. Αναφερόμαστε πολύ συχνά στο θέμα της επαν... Ξέρουμε όμω τι επιπτώσει έχει η κοινωνικο η υλοποίηση αυτού του τεράστιου προγράμματο. Εγώ έχω κάποια στοιχεία τα οποία έχω λάβει από πρόσφατε πηγέ. Ο πρόεδρο μου ρώτησε τι γίνεται στην Ιταλία. Έχουμε 12.000 πρόσφυγε οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη. 31 Δεκεμβρίου ήταν η εκπνοή τη τελευταία προθεσμίας για την υποδοχή τους. Ε, δόθηκε παράταση για 60 ημέρε. επομένως αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δήλωσε ήδη στις τοπικές αρχές ότι θα δοθεί κατά κεφαλήν 400 ευρώ που αν το πολλαπλασιάσουμε με 12.000 έχουμε σημαντικό ποσό για να διευκολύνουμε την ε, εγκατάστασή τους. Και εδώ εγώ αναρωτιέμαι πώς, και σας το λέει και ένας άνθρωπος που δεν είναι και ενθουσιασμένος με τη μαζική μετανάστευση, πώς μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην κοινωνία με 400 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα προβλήματα. Και φτάνω και στο συμπέρασμά μου. Η δέσμη των μέτρων ε, και μας είπε και η κυρία Βάλστρομ η Επίτροπος και εδώ μια και σας μίλησα για υποκριτησία πρέπει να σας το πω γιατί στα θέματα του ασύλου δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς που τότε εκπροσωπούσαμε ε, την αντίθετη θέση ακούσαμε επικρίσεις από μια Επίτροπο η οποία μας έλεγε ότι δεν υποδεχόμαστε και δεν φροντίζουμε αρκετά ε, τους ανθρώπους που έρχονται. Εγώ τότε είπα στον επίτροπο αυτό που δεν θα κατονομάσω ότι στη χώρα τα απαγορεύονται όλα αυτά τα πράγματα και επομένως καταλαβαίνετε πόση υποκρισία υπάρχει. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε η νομοθεσία να μην δώσει δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερες παραβιάσεις και να μην ανοίξουν τα σύνορά μου σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας. Ε, πέραν της περίπτωσης της Σουηδίας, το θέμα τέθηκε και στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στο Δουβλίνο προσφάτω, όπου συζητήθηκε με τον ε, Πρωθυπουργό της Σερβίας, τον κύριο Ντάτσι, διότι εξακολουθεί να εμένει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα ε, με τη Σερβία. Να θέσουμε το εξή ερώτημα λοιπόν. Αρκούν ε, όλες αυτές οι διατάξεις για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις επικίνδυνες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν ε, επειδή δεν τηρείται σωστά η, το ιερό δικαίωμα του ασύλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μποργέτσιο. Λοιπόν. Νομίζω ότι κάπως μακρηγορήσαμε με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, αλλά ξέρετε ο, και το ακούσατε από σήμερα το πρωί ότι πρόκειται για ένα φάκελο πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τις διαφόρες απόψεις, προσεγγίσεις και αναλύσεις. Δεδομένου ότι μίλησε ο συνήγορος του διαβόλου, για συνήγορο του διαβόλου, ο κύριος Μποργέζη, περιμένουμε από εσά να είστε πραγματικά αυτοί που θα κάνετε ερωτήσεις, θα κάνετε σχόλια, όχι μόνο να παρετείτε ερωτήσεις. Αν θέλει καποιο από εσά να κάνει ένα σχόλιο μετά από αυτά που άκουσε από διάφορε παρεμβάσεις των ε, Ευρωβουλευτών, είναι καλοδεχούμενος. Και πρέπει να πω ότι σα ανακαλύπτουμε εμείς. Και εμείς και οι Ευρωβουλευτές. Γι' αυτό να πείτε, σα παρακαλώ, ο καθένα το όνομά του και το μέσο για το οποίο εργάζεται. Παρακαλώ, ποιος θέλει να κάνει την πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Μαριάν Μενιέ, της γαλλικής εφημερίδας Λακχουά. Θα ήθελα να επανέλθω στα ανήλικα μόνα παιδιά. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε την παρούσα νομοθεσία και με ποιο τρόπο η προβλεπόμενη καινούργια νομοθεσία θα βελτιώσει την κατάστασή τους. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πώς θα είναι καλύτερη με το νέο σύστημα η κατάσταση για ένα συνόδευτο ανήλικο παιδί. Βασικά θα έχουμε πιο σαφείς κανόνες. Πρόσβαση στην ενημέρωση. Πρόσβαση σε διερμηνής και μετάφραση. Πληροφορίες ε, που ώρες-ώρες θεωρούμε δεδομένους. Δηλαδή ότι κάποιο παιδί σε κάποια χώρα θα καταλάβει την γλώσσα. Τώρα όμως υπάρχουν πρόνοιες για όλους. Κυρίως όταν πρόκειται για ασυνόδευτο παιδί που έχει το δικαίωμα, όπως είπα, να επανενωθεί με την οικογένειά του, τη μητέρα του, τον πατέρα του, τα αδέλφια του, θείους, θείες, παππούδες, γιαγιάδες, σε άλλη χώρα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα κάνει την κατάσταση πολύ καλύτερη για ένα νέο άτομο, για ένα παιδί και θα είναι και ευκολότερο να χειριστούν την κατάσταση και τα κράτη-μέλη. Θα είναι λοιπόν προς το καλύτερο ε, ένα μέλος της οικογένειας να αναλάβει, να μεγαλώσει, να αναθρέψει ένα παιδί παρά να χρειαστεί να ε, επιληφθεί η κοινωνία. Αυτά λοιπόν είναι τα πάρα πολύ καλά πράγματα που αφορούν τα ανήλικα παιδιά. Και υπάρχει βεβαίως και νομική βοήθεια. Κάποιος ο οποίος ε, θα οριστεί για να φροντίσει το παιδί. Όλες οι διαδικασίες είναι καλύτερες και μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. κύριος Κύρκο, θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλά έγιναν σε πολλούς τομείς για να εξασφαλίσουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι την χάνουν τη κατάλληλη μεταχείριση. Και τα παιδιά, καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είναι και ε, θύματα εμπορίας ο, πολύ περισσότερο από το παρελθόν και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Και βεβαίω θα πρέπει να δούμε με απόλυτη ερμηνεία τι εννοούμε όταν λέμε ανήλικο. Τι είναι παιδί, μέχρι ποιο ηλικία θεωρείται ένα παιδί, παιδί ανάλογα με την νομοθεσία και τη χώρα. Πολλές φορές ε, υπάρχει σύγχυση και πρέπει κάτι να κάνουμε για να υπάρχει πλήρης ε, ε, διαφάνεια για να μπορέσουμε να προστατεύουμε τα παιδιά. Ο κύριος Ιδάλγο. Αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια συζητήσεων για το θέμα της οικογενειακής επανένωσης και των ανηλίκων έγιναν εκτεταμένες, πολύ εκτεταμένες συζητήσεις και αντιφατικές ε, ε, προτάσεις ε, στο σχετικό πακέτο. Όσον αφορά πρώτα απ' όλα την έννοια του τι είναι η οικογένεια, η στενότερη έννοια, η ευρύτερη έννοια και άλλα θέματα. Δεν είναι παρούσα, αλλά θα μιλήσω υπέρ της Jean Lambert που δεν είναι στην ομάδα μου αλλά πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια πολέμησε πάρα πολύ για να ε, ξεκαθαριστεί η κατάσταση σε σχέση με το θέμα που θέσατε εσείς η εκπρόσωπος της Λακρουά ώστε να διευρυνθεί η έννοια της οικογένειας δηλαδή το αν έχουμε να κάνουμε με την ε, νομοθεσία, με τις ε, παραδόσεις, ε, με το τι σημαίνει για κάποια κοινωνία κοινωνία, θα πρέπει να δώσει μια ευρύτατη έννοια, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Διότι πολλές φορές πρέπει να πω στην Ευρώπη είναι πολύ κοινική η θέση μας. Μιλάμε πάρα πολύ για την οικογένεια και την ώρα της αλήθειας τι χτυπάμε την οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν όταν έχουμε πραγματικά σημαντικές περιπτώσεις επανένωσης οικογενειακής, να κινητοποιήσουμε όλα όσα ξέρουμε για την σημασία της οικογένειας από τη θρησκεία για να βοηθήσουν την οικογένεια. Ο κύριος Ταβάρες. Στην περίπτωση των ε, προσφύγων που είναι σε λίστες αναμονής για επανεγκατάσταση, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου χορήγηση, Ασύλου, το οποίο αλλάξαμε και τροπολογήσαμε εμείς το τέλος της Δενικής Προεδρίας, προβλέπει προτεραιότητες για κάποιες κατηγορίες προσφύγων που πρέπει να φροντίσουμε. Μίλησα για 5.000 πρόσφυγες στην Ευρώπη και θέλουμε στα πλαίσια των ΜΚΟ που εργάζονται σε τέτοιου είδους θέματα κατάσταση και των πολιτικών στήριξης και συμφωνήσαμε να φτάσουμε το 2020 σε μετεγκατάσταση και αποκατάσταση 20.000 προσφύγων. Σύμφωνα με κατάλογο, έτσι όπως προβλέπετε στον ε, τροποποιημένο αυτό κανονισμό προσφύγων, επαναλαμβάνω, που είναι κατά προτεραιότητα αυτοί που ήταν θύματα ε, σεξουαλικής ε, βίας, σωματικής βίας, θύματα βασανισμών, παιδιά, ανήλικες, άτομα τα οποία επέστησαν κάποια απειλή και ένα από τα κριτήρια αυτής της λίστας προτεραιότητας είναι το κριτήριο του ασυνόδευτου, του μόνου ανήλικου παιδιού, οπότε θα πρέπει να γίνει με την κατάσταση και αποκατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς συμφέρον του παιδιού, διότι ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε περιπτώσεις ανηλίκων όπου μπορούν να τύχουν της υποστήριξης της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ ή κάποιο άλλο φορέα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κριτήρια που θα ακολουθηθεί. διότι υπάρχουν μόνα τα παιδιά που πρέπει να πάνε σε μια τρίτη χώρα την οποία δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν κανένα, δεν ξέρουν ακριβώς τα συμβεί. Πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για να ξέρουμε πάντα ποιο είναι το καλύτερο συμφέρον των παιδιών το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Ε, επιστροφής των προφύγων και των κριτηρίων που ακολουθούνται και η επανεγκατάσταση στην Ευρώπη, θέματα για τα οποία επίσης εργάζεται και ο συνάδελφος Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, όλες οι δραστηριότητες αυτές θα τεθούν από κοινού στο νέο Ταμείο Μετανάστευσης Ασύλου με εισηγήτρια την κυρία Σιλβί Γκυγιόμ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται η κυρία Γκυγιόμ με το Συμβούλιο. Και βεβαίως θα εξαρτηθούν και πολλά από αυτές τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου για να δούμε ποιες αλλαγές θα γίνουν και ποιες βελτιώσεις ώστε τα άτομα που αναφέρατε να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Ευχαριστώ. Εδώ μπροστά μια κυρία θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Bon, ε, Vous êtes... Το μικρόφωνο να ανοίξετε παρακαλώ. Μαρία Σιντηροπούλου from Sky TV Greece. Um, uh, I don't know if you're aware. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι συνέβη πριν από δύο εβδομάδες στην Ελλάδα με δύο μετανάστες που διέφυγαν από ένα κέντρο φύλαξη στην Ελλάδα εξαιτία των απάνθρωπων συνθήκων που επικρατούσαν. Τους αθώσε το ελληνικό δικαστήριο για αυτό που έκαναν. Έπρεπε να διαφύγουν εξαιτίας αυτών των απάνθρωπων συνθήκων, αλλά θα ήθελα να σας ερωτήσω δεδομένου ότι έχει υποστεί πολλές οικονομικές κυρώσεις για αυτά τα θέματα η Ελλάδα, πιστεύετε ότι αρκούν ή υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προβλεφθούν νέα συστήματα εποπτείας, πιο συστηματική έλεγχη για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την ερώτηση. Όσον αφορά την κράτηση, θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σαφής. κράτηση για τον απλό και μόνο λόγο ότι είσαι τον ασύλου όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Ιταλία και έχω, τα, τα έχω δει όλα αυτά τα κέντρα κράτησης δεν θα επιτρέπεται πλέον. Απαγορεύεται αυστηρά η κράτηση ατόμων που κάνουν αίτηση ασύλου σε περιπτώσεις ε, του κανονισμού του Διβλίνου. Και πάλι μπορεί να υπάρξει κράτηση, αλλά μέχρι τρεις μήνες, το αργότερο τρεις μήνες. Αλλά εγώ προσωπικώς έχω γνωρίσει ετούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν ε, κρατηθεί στην Ελλάδα και στην Ιταλία για μήνες και χρόνια. Για τον απλό και μόνο λόγο γιατί ε, ζητούν διεθνή προστασία στην Ευρώπη και αυτό φυσικά είναι απαράδεκτο και δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θέσατε αυτή την ερώτηση, διότι η κράτηση είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε και δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι δεν είναι αντάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωση στον 21ο αιώνα να συμπεριφέρεται στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τώρα τι κυρώσει. Δεν υπάρχουν κυρώσει, αλλά Αυτό το οποίο είναι ουσιαστικό για όλο το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου είναι κάθε κράτος μέλος να είναι αντάξιο των κανόνων αυτών, να φανεί στο ύψο των περιστάσεων, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη. Ότι εσεί θα αναλάβετε τι ευθύνε σα, εμεί θα αναλάβουμε τι δικέ μα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου θα ε, συμπεριφέρονται στου ανθρώπου επί ίση όρη και δεν θα υπάρχει διαφορά αν ε, κάποιο είναι. Ε, ετών άσυλο και καταλήξει στις ακτές της Ελλάδος ε, ή πάει στη Σουηδία ή στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Είμαστε μια ένωση που βασίζεται σε κοινέ αρχές και θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί το σύστημα. Επίσης, ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι το σύστημα αυτό δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της καθυστέρησης και του προβλήματος που υπάρχει στις Σικελία στην Ελλάδα αλλά δεν θα επιτρέψει να πέσουμε στην ίδια παγίδα σε άλλα κρατημέλη ε, και να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης, μπορείτε να μιλήσετε και ελληνικά. Υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά. Επειδή ετέθη η ερώτηση στα αγγλικά, θα απαντήσω αγγλικά. Yes, I also want to thank Mrs. for this question. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Σιδηροπούλου για την ερώτηση διότι θέτει όλα τα ζητήματα τα οποία ανέφερα προηγουμένως, το θέμα της αλληλεγγύης, ας πούμε. Πρέπει βεβαίως να πω ότι αυτές οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι πολύ χρήσιμες για μας, διότι δείχνουν τι θα πρέπει να κάνουμε και όχι τι έχει γίνει μέχρι τούδε. Πρέπει να πω ότι η κατάσταση στην Ελλάδα διαφέρει ιδιαίτερα από το πώς ήταν όταν ε, ε, λήφθησαν υπόψη συγκεκριμένε προποθέσει στην Ελλάδα. Εμεί ω Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων ε, κάναμε αρκετέ αποστελέ στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη ήταν πριν από δύο μήνε και είδα πολύ μεγάλε αλλαγέ. Όχι γιατί επιβλήθησαν κυρώσει και σε αυτό θέλω να καταλήξω, αλλά γιατί επεδείχθη αλληλεγγύη. Και θεωρώ ότι οι κυρώσει θα πρέπει να είναι ίστατη λύση θα είναι πολύ καλύτερο να επιδείξουμε αλληλεγγύη, να συνδράμουμε μια χώρα σαν την Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να υπερκεράσει τι δυσκολίες τη. Και τα εργαλεία στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένω έχουν τεθεί σε πρακτική εφαρμογή. Για παράδειγμα, η ΆΣΟ ε, βοήθησε ιδιαίτερα διότι εκπαίδευσε τι ελληνικέ αρχέ για το τι να κάνουν με τι αιτήσει, με τι συνθήκε κράτηση. Και ο Frontex έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, διότι σταμάτησε την εισρωή μεταναστών στην περιοχή του Εύρου. Επομένως, θεωρώ συμπερασματικά ότι η παρακολούθηση είναι καλή. Με τις κυρώσεις δεν συμφωνώ, αλλά η αλληλεγγύη είναι ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδείξει στην πράξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μποργκέτσιο. Πολύ ε, συνοπτικά θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το γεγονός ότι στο παρελθόν πριν από την έγκριση της συγκεκριμένη διάταξης υπήρχαν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβαινε σε κάποιες χώρες αυτό διότι δεν ήξεραν ποιος είναι αυτός ο οποίος καταθέτει αίτηση ασύλου και σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες φτάνουν χωρίς έγγραφα και είναι πολύ δύσκολο να ε, τους βρούμε. Δεν υπάρχει και συνεργασία από τις αρχές της χώρας καταγωγής και επομένως υπάρχει ανάγκη για την ασφάλεια όλων και για τους υπολείπους που έχουν δικαιώματα πρόσφυγα ε, να ε, κρατούνται. Και θεωρώ από αυτή την άποψη ότι η Eurodac συνεισφέρει διότι μπορούμε να διευκολύνουμε πολύ την ε, ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων και έτσι θα υπάρχει μικρότερη ανάγκη για την ανάγκη αυτή που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Ο κύριος Σταβάρες. Συγγνώμη, θα ήθελα να πω το εξή. Όταν είπα απάνθρωπες συνθήκες, εννοούσα απάνθρωπες συνθήκες. Οι εγκληματίες ε, στην Ελλάδα έχουν ε, καλύτερες συνθήκες στις φυλακές. Σε αυτό αναφερόμουν. Όταν δεν γνωρίζουμε ποιος έρχεται, δεν σημαίνει ότι τον, ε, του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι χειρότερος από εγκληματίες. Αυτό ήταν αυτό το οποίο ήθελα να πω. Ο κύριος Σταβάρες. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Να πω κάτι. διότι συμφωνώ απόλυτα με κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν από τους ε, συναδέλφους, από την κυρία Γουίκστρομ και κάποια από τα οποία είπε ο Νίκος Καλό είναι όμως να σταθούμε σε κάτι που είπε η Σεσίλια στην ομιλία της. Εάν οι πολιτικές αυτές διέπονται από την αλληλεγγύη ή από τις ε, μεταναστευτικές ροές. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Συστηματικά όταν ασχολούμαστε με αρκετά τέτοια θέματα, ε, αρκετοί εισηγητές και εγώ και οι άλλοι επιλέγουμε ως νομική βάση, τη νομική βάση που μας παρουσιάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως, το άρθρο 80. Το άρθρο 80 αφορά την αλληλεγγύη, όχι μόνο αλληλεγγύη προς τον πρόσφυγα, αλλά και αλληλεγγύη ε, υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να επιδεικνύουν αλληλεγγύη ο ένας τον άλλον. Πρέπει δηλαδή να βοηθούν ο ένας τον άλλον για να υπάρχουν καλά συστήματα ασύλου. Υπ' αυτή την έννοια οι κυρώσει δεν έχουν αποτέλεσμα. Το Συμβούλιο όμως την αλλάζει πάντα τη νομική βάση και πηγαίνει στο άρθρο 76G που αφορά μόνο τις μεταναστευτικέ ροές. Δηλαδή κάνουμε διαχείριση μεταναστευτικών ροών διότι δεν θέλουν να πληρώνει ο ένα για τον άλλον. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με κατάλληλου Ευρωπαϊκού μηχανισμού, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ίδιου πόρου κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό σημαίνει ότι αρκετά κράτη-μέλη που αυτή τη στιγμή έχουν πληθώρα ενστάσεων, όταν δεν θα πρέπει να τα πληρώσουν, θα σταματήσουν τι ε, ενστάσει του και θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν προσπαθούν ε, σώνη και καλά να φτάσουν στην Ελλάδα ή στη Μάλτα ή στην Κύπρο, προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και υπ' αυτή την έννοια το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Ο κύριο Στις παρατηρήσεις που έδωσα προηγουμένως, σας είπα στο τέλος, σας ανέφερα κάποιο παράδειγμα. Πρέπει να πω ότι δεν είχαν ούτε και σωστά στρώματα να κοιμηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις ε, οι πρόσφυγε. Ίσως και στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό θέλω να μιλήσαμε για αλληλεγγύη. Αλλά θα πρέπει να έχει αυστηρή γραμμή πλεύσης η Κομισιό με τις χώρες που δεν ε, ε, δίνουν και τα απαραίτητα βασικά εχέγγυα αξιοπρεπίας τους ε, υποψήφιους πρόσφυγες. Όποια και κυβέρνηση, σε όποια χώρα και να είναι, εάν δεν προσφέρει minimum standards, τι κάνει. Διότι η κατάσταση για κάποια άτομα έχει ως εξής. Ακόμη είναι σε κατάσταση αναμονής. Για πρέπει να τους μεταχειρίζεται κανεί χειρότερα από ότι έναν ε, εθνικό εγκληματία. Θα πρέπει λοιπόν να, ε, η Κομισιόν να πει στα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν. Πάρα πολύ καλά τα είπε, Τίμωθη. Δηλαδή, να ενεργήσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάτι σωστό. Τώρα, είναι επανέλθω στην αλληλεγγύη και στο άρθρο 8 των ε, ε, συνθήκων. Θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική για θέματα αλληλεγγύης και να είναι δεσμευτική για όλους. Και θα ήθελα να προσθέσω στην ε, πράξη η αλληλεγγύη για τη Σουηδία τι σημαίνει, ότι περισσότερα από 40 άτομα πήγανε στην Ελλάδα ώστε να αρχίσει να λειτουργεί κάπως το σύστημα ασύλου, διότι η αλήθεια είναι στην Ελλάδα όχι ότι έχει καταρρεύσει όπως είδαμε σε κάποιες εφημερίδες, αλλά ποτέ δεν δημιουργήθηκε σε πρώτη φάση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση τώρα, ότι τέθηκε σε κίνηση, σε λειτουργία και φαίνεται ότι λειτουργεί και βεβαίως θα υπάρχει αποπτία και παρακολούθηση, αλλά η αλληλεγγύα τι σημαίνει, ότι θα πρέπει επίσης να προσφέρουμε και τους ανθρώπινους κατάλληλους πόρους για να κάνουμε την πολιτική. Ε, πολύ συνοπτικά θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Σκεφτείτε την περίπτωση της Λαμπεντούζα. Ε, είχαμε αφήξεις ε, και φυσικά υπήρχε και παρουσία ατόμων που είχαν δικαίωμα σε καθεστώς πρόσφυγα, ε, αλλά είχαμε όλες αυτές τις οριδών αφέξεις που ήταν η Ευρώπη. Υπήρχε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στη Λαμπεντούζα. Υπήρχε παρουσία νομική, παρουσία θεσμική. Όχι. Και εν μέσω κατεπίγουσας κατάστασης είχαμε ακόμα και μαγνητοσκόπηση δύο υπαλλήλων που ήρθαν ευσπεσμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γυρνούσαν στους δρόμους της Λαμπεντούζα και νομίζω ότι ε, σε ένα μπαρ είχαν στήσει ένα γραφείο και δουλεύανε. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε καμιά δομή να τους φιλοξενήσει. Ενώ λοιπόν οι επίσημες τοπικές και κυβερνητικές δομές στην Ιταλία δραστηριοποιούνταν πλήρως και έκαναν ε, με όλες τις δυσκολίες και με όλα τα ελαττώματα στα οποία δεν θα σταθώ αυτή τη στιγμή όλη τη δουλειά δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στα κράτη-μέλη κάθε φορά. Πολύ συχνά όταν υπάρχει έλλειψη συντονισμού ή αναπάρκεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλο το βάρος πέφτει σε χώρες ε, που έχουν εξωτερικά σύνολα, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο ακόμα και αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Ένα σύντομο σχόλιο για τη Λαμπεντούζα δεν μπορώ να μην το πω, διότι πρέπει να το πω οπωσδήποτε. Πρόκειται για ένα τεράστιο ευρωπαϊκό σκάνδαλο. Το γεγονός ότι το λιμάνι της Λαμπεντούζα θεωρήθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση ως ε, ε, επικίνδυνος λιμένας, αλλά όχι εν γέννη επικίνδυνο για τους ετούντες άτυσίλο και τους πρόσφυγες, αλλά όχι επικίνδυνο για τους τουρίστες και τους αλλοίς, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη και αυτό είναι ε, απαράδεκτο. Χάρη σε μια νέα απόφαση η οποία λήφθη από την Ιταλική κυβέρνηση και χάρη στο νέο δήμαρχο, στη νέα δήμαρχο μάλλον, μια γυναίκα η οποία κατάγεται από την περιοχή της Λαμπεντούζα, άλλαξε η νοοτροπία. Αλλά πρόκειται για ένα τεράστιο ευρωπαϊκό σκάνδαλο, το γεγονός ότι το λιμάνι αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, έπρεπε, είχε το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί δεν πρέπει να ξανασυμβεί σε καμία περίπτωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την υπενθύμηση κυρία Βίκστρομ. Μία ερώτηση από την κυρία Μελίτα Σούνιτς από το Γραφείο των Βρυξελών ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να μην είναι δική μου δουλειά γιατί αυτό είναι ένα σεμινάριο για τους δημοσιογράφους, αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι το οποίο ουσιαστικά διέπει όλες τις δηλώσεις του κυρίου Μποργέτσιο. Όποιος τις δηλώσεις του εξακολουθεί ή μάλλον το θέσω αλλιώ. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Εγώ ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών ουσιαστικά προασπίζομαι την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε έναν Ευρωβουλευτή, αλλά θα το κάνω στις δηλώσεις σας συνεχώς ε, αναμειγνύεται διάφορα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα την περίπτωση του ασύλου και των ατόμων που ζητούν προστασία, την οικονομική μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, την ε, διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και κατηγορείται την νομοθεσία για το άσυλο διότι δεν βοηθά όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά τα φαινόμενα, κατά την άποψή μου, έχουν σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, είναι αλληλένδετα. Αλλά η νομοθεσία για το άσυλο στόχο έχει να καθορίσει σε ατομικό επίπεδο τον άνθρωπο που θα έρθει στα σύνορα και θα πει ότι εγώ ζητώ άσυλο. Η νομοθεσία ασύλου θα φροντίσει να, να σε μεταχειριστούν σωστά, να σου συμπεριφερθούν σωστά, να μπορέσουν να δούνε οι αρχές αν όντω ε, χρειάζεσαι άσυλο και προστασία ή όχι και υπάρχει και ε, ένας βαθμός αμοιβαίας ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ασύλου. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορείς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ασύλου διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχει θεσπιστεί γι' αυτό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να επιληθούν με πολιτικό τρόπο. Όλοι γνωρίζουν ότι αν θέλει να σταματήσει η ροή σύρων προσφύγων πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Συρία και η νομοθεσία για το άσυλο δεν υπεύθυνη γι' αυτό. Εάν ε, θέλει κάποιος να ασχοληθεί με τη μετανάστευση των Ρωμά που γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ε, σε άλλες χώρες ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός, ε, οι Ρωμά πηγαίνουν και ζητούν άσυλο στην Καναδά για παράδειγμα, ε, δεν μπορούμε να την αποκαλούμε αυτήν πολιτική αριβεντέρτσι Ρώμα, κλείνουμε τι πόρτε και αρνούμαστε τι θεωρήσει και λέμε δεν μα ενδιαφέρει η φτώχεια σα, δεν μα ενδιαφέρουν πολιτική περιθεριοποίησή σα και κοινωνική περιθεριοποίησή σα, δεν σα θέλουμε εδώ. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα και η πολιτική μετανάστευση και πάλι δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα του ετούντο άσυλο, αλλά είναι η περίπλοκη κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση. Και εδώ λοιπόν εγώ Σα λέω ότι είναι καλό το γεγονό ότι υπάρχει ένα κοινό σύνολο κανόνων πλέον. Πόρο απέχουμε από την πλήρη αναρμόνιση τη πολιτική ασύλου και μετανάστευση, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νόμους που έχουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεμονωμένες αιτήσει ασύλου και να καθορίσουμε άλλους κανόνες που αφορούν την εμπορία, τη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα, γιατί ε, εκεί πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Επειδή η ερώτηση ετέθη προς τον κύριο Μποργέτσιο, να του δώσω το λόγο. Εγώ δεν θα σας πω την προσωπική μου άποψη, διότι είναι γνωστό τη σπάση ότι ο ΙΕ, ο, ο οποίος παρενέβη σε αυτή την περίπτωση, θεώρησε ότι προσβάλλεται επειδή θέτω συνεχώς ερωτήσεις και προς το Ιταλικό Κοινοβούλιο, διότι με σκανδαλίζει το γεγονός ότι είναι συνεχώς υπάλληλοι παρόντε σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, οι οποίοι πρέπει να ασχολούνται με πιο αποτελεσματικό τρόπο με αυτές τις περιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη, συζητήθηκε το θέμα του λιμανιού της Λαμπεντούζα. Τι έκανε ο ΙΕ για να επισημάνει το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της ε, συνεχούς ροής μετανάστευσης εις βάρος ενός φτωχού πληθυσμού ε, των ε, αλλιέων και των εργαζομένων στη Λαμπεντούζα που δεν μπορούσαν να κάνουν καν τη δουλειά τους διότι το λιμάνι ήταν γεμάτο από εκατοντάδες ε, βάρκες εμπόρων ανθρώπων και παράνομων μεταναστών. Αναφέρεστε επίσης στην εφαρμογή των ιερών μέτρων ε, για, τα, για το άσυλο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι έμποροι ανθρώπων για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις και επαναλαμβάνω οι υπάλληλοι τους παίρνουν υπέρογους μισθούν και ζουν μέσα στην πολυτέλεια και δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το να καταγγείλουν και να ε, υποδείξουν κανόνες που θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις και στις διεθνείς διεθνείς οργανώσεις να ε, σταματήσουν την εμπορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, στη Λαμπεντούζα θα μπορούσε να ε, είχε υπάρξει ένας ε, σημαντικός χώρος και να γίνει μια παρέμβαση για να επιληθεί κάτι τουλάχιστον. Παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Ωραία, έχουμε δύο ερωτήσεις. Συγγνώμη, διότι πρέπει να συνεχίσουμε. Μπορείτε να κάνετε σχόλια λίγο αργότερα. Αλλιώ ε, δεν θα μπορέσουμε να. θα έχουμε ένα πέρα δόθε και θέλουν να λάβουμε το λόγο και οι δημοσιογράφοι. Εσεί και στη συνέχεια ο κύριο στο βάθο. I'll speak Greek, okay? Thank you. Ah, you know Greek. Oh. Κατάλαβε Okay. Ε, το όνομά μου είναι Δελιθανάση από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ε, θα ήθελα να πω στον κύριο Μποργκέζη ότι με ανάλογα επιχειρήματα θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά και για τον θόκο τον οποίο ο ίδιος κατέχει. Θα μπορούσε να μιλήσει για πολυτελούς, ε, για ευρωβουλευτές οι οποίοι διαβιούν ε, με τρόπο που δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία και δεν κατανοούν τι ακριβώς συμβαίνει και επί τη ευκαιρία, επειδή το νιώθω πλέον σε εσωτερική ανάγκη ως πολίτης, να τον ρωτήσω αν θεωρεί λοιπόν, ε, λέει, είπε πριν ότι με 400 ευρώ ποιος ε, αλλοδαπός ή ε, πρόσφυγας θα μπορούσε να ζήσει εδώ χωρίς να συνιστά κίνδυνο. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω αν θεωρεί λοιπόν ότι συνιστά κίνδυνο, συνιστού... θα σας πω ακριβώς... Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα ε, με τη μετάφραση, είπε ο κύριο Μποργκέτσο. Εγώ είπα ότι είναι αδιανόητο να μπορούμε να εντάξουμε κάποιον με 400 ευρώ. Το αντίθετο είπα. Συγγνώμη κύριε Μποργκέτσο. Είπατε ακριβώ πώ μπορεί ένα άνθρωπο να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία με 400 ευρώ. Σωστά. Α, σε la αλλά είναι πάρα. It's not the proper. It's okay, it's okay. Okay. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέτει ζητήματα τα οποία, αν μου επιτρέπετε, επιχειρηματά του τα θεωρώ έολα. Με την ίδια έννοια θα λέγαμε πώς μπορεί ένας Ευρωπαίος ε, να ενταχθεί, να παραμείνει ενταγμένος στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία με 400 ευρώ. Okay. Τέλος πάντων, θα ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ε, το οποίο έχει να κάνει, γιατί το θέμα των συνθηκών υποδοχής το εξαντλήσατε, το οποίο έχει να κάνει με το Δουβλίνο. Και ήθελα να ρωτήσω το εξή, επειδή το θέμα Δουβλίνο για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο ή κάποιε χώρε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης είχε διατυπωθεί ποτέ κάποια σκέψη να υπάρχουν γραφεία χωρών ε, όπως π.χ. της ε, Σουηδίας, την οποία αντιπροσωπεύει η κυρία βιξτρομ που θα φρόντιζε για λόγους ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ευρωπαϊκού ανθρωπιστικού δικαίου ανήλικους ή άλλους ευάλωτες ομάδες, να τους διευκόλυνε ώστε άμεσα να μεθεγκατίστανται σε άλλες χώρες και να μην περνούν μέσα από την ταλαιπωρία της ελληνικής διαδικασίας που είναι εξαιρετικά τραυματική και το ξέρετε. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Μασίπ Ιντάλγο, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Να σας πω ότι πραγματικά συγκινούμε ότι ακούμε μία εκπρόσωπο του ΟΗΕ σήμερα να μιλά εδώ, σε ένα τέτοιο χώρο, γιατί πρέπει να σας πω ότι η πολιτική μου εμπειρία, που είναι εμπειρία πολλών ετών, αλλά και ως Ευρωβουλευτής από το 2004 εδώ, έχω δει ότι η Πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες είναι υποδειγματικός οργανισμός υποδειγματικός ε, και λόγω των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για κάθε έναν από τους εργαζομένους τους, άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στην υπατιαρμοστία. Και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ χειρότερος χωρίς ε, την υπατιαρμοστία για τις πρόσφυγες. Έχω επισκεφθεί πάρα πολλά στρατόπεδα προσφύγων ε, και στην κοντινή περιοχή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αλήθεια είναι ότι πάντα ε, συναντούσα την είπατε αρμοστία και ποτέ δεν είδα σύμπτωμα προνομίων και πολυτέλειας. Πάντα έχω δει απόλυτη υπευθυνότητα. Ε, θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που προασπίζονται τις οδηγίες ε, που κάνουμε και αποτελούν παράδειγμα για μας και το μόνο που με λυπεί είναι ότι η έκθεσή μου δεν είναι όσο καλή θα ήθελα να ήταν διότι εγώ είχα γράψει μια προηγούμενη έκθεση που εγκρίθηκε εδώ στις Βρυξέλλες στο Κοινοβούλιο το 2000 κάτι στην τελευταία ημέρα της προηγούμενης θητείας που ήταν καλύτερη από την έκθεση που έχουμε τώρα. Αλλά τι συμβαίνει. Μετά κάποιες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και οι κυβερνήσεις που αναφέρεται προηγουμένως, δεν έδιναν ε, ε, το πράσινο φως για να προχωρήσει. Εγώ στα νιάτα μου ήμουν επαναστάτης, αλλά τώρα πια δεν είμαι είμαι πρακτικός άνθρωπος και προσπάθησα να βρω μια λύση για όλες αυτές τις υποθέσεις. Και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μια λύση που είναι σχετικά καλή και όπως σας έλεγα προηγουμένως πρέπει, όπως είπε και η κυρία Γουίξτρομ προηγουμένως, δεν πρέπει ποτέ να δεχτούμε ένα άνθρωπο που έρχεται στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που κάνει η Ευρώπη είναι να τον θέτει υποκράτηση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πέντε λόγοι συντρέχουν για την κράτηση βάσει της οδηγίας, πέντε μόνο, και ε, το οποίο για μένα και αυτό θα έπρεπε να το επικρίνουμε, αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να περάσει αυτή η υπόθεση. Δεν πρέπει να κρατείται κανείς. Και παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να προσφύγει απευθεία ε, στα δικαστήρια, υπάρχει όμως η περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος ε, που είχαμε στην Ελλάδα και θα μπορούσαμε να έχουμε και στο παρελθόν, να σας πω ότι εγώ είμαι νομικός. Και δυστυχώ αυτό δεν είναι πλέον δίκαιο θεσπισμένο, διότι μας λείπει ένα τελευταίο στάδιο κάποιων μηνών εδώ στο Κοινοβούλιο μέχρι να εγκριθεί οριστικά η νομοθεσία και να γίνει αποδεκτή από τις κυβερνήσει. Είμαι βέβαιος όμως ότι κάποιο δικηγόρος, καλύτερος από μένα, παντού στην Ευρώπη θα μπορέσει να ζητήσει να εφαρμόζεται στην οδηγία αυτό, αυτό το οποίο αποκαλούμε νόμος ενισχύ, λέχε φερέντα, για τους Ευρωπαίους και τους Ευρωπαίους νομοθήτες ε, υπάρχει αυτή η διαδικασία και θα πρέπει να το ζητούμε και κανείς δεν θα πρέπει να κρατείται στην Ευρώπη παρά μόνο για αυτούς τους τέσσερις λόγους που αναφέρονται στην οδηγία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύρκοφ θέλει να σχολιάσει. Κοιτάξτε, να πω το εξή. Όλη αυτή η συζήτηση για την Ελλάδα και τις δύσκολες συνθήκες και το καθεξής. Βεβαίως και θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη όταν μπορούμε, όταν αντιμετωπίζουν ε, ε, δυσκολίες για να υποδεχθούν όλους τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα. Αλλά η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αφήξεων, αιτήσει ασύλου και επισήμως ε, δέχονται μερικές εκατοντάδες. Ενώ ταυτόχρονα η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες ε, υποδέχονται χιλιάδες ε, πρόσφυγες στο ίδιο διάστημα και θα πρέπει να το δούμε και το θέμα λίγο στη σωστή του διάσταση πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί για τι προποθέσει που ισχύουν για αυτού τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία φτάνουν. Η κυρία Βίξτρομ, για να επανέλθω στην αλληλεγγύη, για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Εγώ δεν μίλησα για στήριξη σε χώρες. Αναφέρθηκα σε στήριξη προς τους ανθρώπους. Και να επανέλθω στην ερώτησή σας από διαφορετική οπτική γωνία. Εδώ η πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι 17 χώρες συνεισφέρουν και τη μόνο της δεσμεύσεις τους για να θεσπίσουν το σύστημα χορήγησης ασύλου. Και αυτό θα διευκολύνει την πίεση των 10 χωρών που δέχονται περισσότερο από 90% των τον ασύλων. Και η, χώρα, η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες. Αυτή είναι η πραγματική λοιπόν αλληλεγγύη. Δηλαδή, οι χώρες που σχεδόν δεν ικανοποίησαν κανένα αίτημα ασύλου να αποδείξουν τη βούλησή τους και να πούν ότι Όντω είμαστε μέρο του κοινού συστήματο χωρί ασύλου στην Ευρώπη, είμαστε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα όπω το εφαρμόζουν τη χωρί ασύλου και οι άλλε χώρε μέλη. Ευχαριστώ. Μια στιγμή. Παρακαλώ. Με τη σειρά ο καθένας. Γεια σας. Είμαι ο Γιάνκοβιτς από την ε, ε Σλοβενία, προδιοφωνικό σταθμό. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μετά από αυτό που ο κύριος Θα Πολλά ελέγχθησαν. απλώ να πω ότι θα πρέπει, παρόλο που κάνετε το ε, σύνδεκο του διαβόλου, να προσέξετε το εξή. Να συνδέετε τους πρόσφυγες με τα θέματα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Πρέπει να σας πω ότι Γνωρίζουμε ότι στην Ιταλία γίνεται και μεγάλη εμπορία ανθρωπίνων ε, όντων. Ε, από την τραγκέτα, όπως είπατε. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι έχουν λοιπόν πολύ αρνητική άποψη για τους ε, πρόσφυγες, δεδομένου ότι διασυνδέουν και την τράγκετα και την εμπορία ανθρωπίνων όντων που κάνουν. Πολλοί όμως από αυτούς τους ε, μετανάστες και πρόσφυγες ασχολούνται ε, και χωρίς να έχουν ε, επίσημα χαρτιά με την καλλιέργεια. Τι προτίθεται να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εγκληματικές οργανώσεις που παρεκκλίνουν από την κοινοτική νομοθεσία και δεν είναι σε θέση να ε, διορθώσουν την κατάσταση ενώ πολλές φορές χρησιμοποιούνται και προς δικό τους όφελος. Αμέτζι από την Media Press στη Γαλλία. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις που αφορούν την γεωγραφική θέση της όλης προβληματικής ε, ε, μετακίνηση των ατόμων και κυρίως των ετούν τον άσυλο. Βλέπουμε από την επικαιρότητα ότι γεωγραφικά οι χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Είναι μια πραγματικότητα σε αυτό το φαινόμενο. Πολύ συχνά βλέπουμε σε αυτές τις χώρες να καταφθάνουν άτομα που ζητούν άσυλο. Το ερώτημά μου είναι πώς χειρίζεται το πρόβλημα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνει υπόψη αυτό το θέμα της επανένωσης των οικογενειών ή μάλλον της αντιμετώπισης των οικογενειών. Διότι όλο και περισσότερο βλέπουμε να φτάνουν μαζικά οικογένειες. Μάνα, πατέρας και παιδιά. Και υπάρχουν χώρες που είναι πιο ευνοϊκές για να δεχθούν ένα παιδί, για να πάει στο σχολείο και από τη στιγμή που πρέπει να έρθει και η οικογένειά του γίνονται πιο σκληρέ. Δεύτερον, μπορούμε να προβλέψουμε, όχι για αύριο, αλλά σε κάποια χρόνια, ότι όπως είπε η Ελληνίδα συνάδελφος, μίλησε για αλληλεγγύη. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε οι ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτούν κάπω την αλληλεγγύη τα πλαίσια της υποδοχής των ατόμων αυτών. Δηλαδή, πώς θα μοιραστούμε τα άτομα αυτά τα οποία είναι σε κατάσταση αναμονής για να γίνει αποδεκτή αίτηση ε, ασύλου. Είναι κάτι το τοπικό αυτό το οποίο λέγω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης ή όχι, είναι κάτι που προβλέψει ότι μπορεί να συμβεί. Πολύ σύντομα, για να απαντήσω το δεύτερο ερώτημα, λέει ο κ. Κύρκο. διότι νομίζω ότι ο Γάλλος δημοσιογράφος θα συνειδητοποιεί ότι η Γαλλία δεν κάνει όχι μόνο αυτά πρέπει να κάνει, αλλά πολύ περισσότερα. Είναι σε πάρα πολύ καλή θέση όσον αφορά το ανθρωπιστικό, ε, την ανθρωπική διάσταση του όλου προβλήματος των προσφύγων. Το δεύτερο ρώτησε, αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να μοιραστούμε τις ευθύνες. Βεβαίως, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά πάντα είχαμε πρόβλημα αυτό το θέμα, διότι οι πρόσφυγες πάνε ε, σε κάποιες χώρες και όχι σε άλλες. Και δεν θέλουν να χειριστούν το θέμα αυτό τόσο ε, θετικά όπως το χειρίζεται η Γαλλία. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ. Κατανοώ τα επιχειρήματά σας για τις μεσογειακές χώρες, για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Το κατανοώ πλήρω και το δέχομαι. Δεν θα πρέπει όμως ως επιχείρημα να το χρησιμοποιούν οι χώρες αυτές για να πούν ακούστε είμαστε πιο ευάλωτες και τα ρεύματα των προσφύγων φτάνουν προς εμάς. Όταν άρχισα σήμερα το απόγευμα σας έδωσα το παράδειγμα των ε, τον άσυλο από το Κωσυφοπαίδιο. Σε ένα χρόνο δεχτήκαμε εμείς 82.000 άτομα στη Σουηδία. Πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη σημερινή Ευρώπη. Δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής. Αν συμβεί κάτι στον Πελαρούς, πού θα πάνε αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες. Στη Λιθουανία, έτσι. Και θα πάνε στην Πολωνία. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι δεν έχουμε ειδικά μέτρα για τις χώρες της Μεσογείου, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα εποπτεύει το γραφείο Ιάσο και θα ελέγχει και την δυνατότητα υποδοχής των ετούντων άσυλο σε όλες τις χώρες μέλη. Και εδώ επίσης έρχεται το 2013 13 ο μηχανισμός έγκαιρη Προειδοποίησης που είναι μια εξαιρετική πρόταση και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή. Διαβάστε αν δεν το έχετε διαβάσει, διότι έτσι επιλύονται όχι μόνο τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά γίνεται προσπάθεια να αποτραπεί και οποιαδήποτε μεγάλη αποτυχία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ε, στο μέλλον ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Έτσι πρέπει να θέσουμε τα πράγματα. Άκουσα, πιστέψτε με, εκατοντάδες επιχειρήματα από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Κύπρο, από τη Μάλτα και από άλλες ε, ε χώρες που είναι στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν να ήθελαν κάτι περισσότερο σαν να έπρεπε να σχεδιαστεί το σύστημα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των χωρών. Αλλά αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα και μιλούμε βεβαίως και για άτομα τα οποία διαφεύγουν από δύσκολες πολιτικές καταστάσεις, από τρίτες χώρες, από, καταστα... χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά μπορούμε να έχουμε και ε, πρόσφυγες και τούντε άσυλο από χώρε στι οποίε έχει υπάρξει μια μεγάλη φυσική καταστροφή και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε χώρα του κόσμου. Όντω χρειαζόμαστε περισσότερε φιλοσοφικέ συζητήσει για τη μετανάστευση για να φτάσουμε σε πραγματιστικέ λύσει. Αλλά έχουμε όντω να κάνουμε με ένα ευρύτατο πρόβλημα. Ρούι Πάρα πολύ σύντομα. Και τώρα θα μιλήσω πορτογαλικά. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση για την οργανωμένη εγκληματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια ειδική επιτροπή αυτή τη στιγμή που εργάζεται σε θέματα ε, ξεπλήματος χρήματος, διαφθοράς και οργανωμένου κλίματος. Πρόκειται για μια ειδική υποεπιτροπή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και συζητώνται εκεί διάφορα μέτρα τα οποία έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα θα κάνουμε συστάσεις στην ε, Επιτροπή ώστε να αρχίσει μετά η Επιτροπή ε, νομοθετικές διαδικασίες. Και τα μέτρα τα οποία συμβουλεύουμε είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο με τα χρήματα τα οποία ε, ανήκουν στη μαφία και έχουν και μπορούμε να ακινητοποιήσουμε ή κέρδη από παράνομο χρήμα, συστάσεις για να πολεμήσουμε την, οικονομική εγκληματικότητα και βεβαίως αυτό είναι και ένα θέμα που απασχολεί πολλά κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ενιαία φορολογική πολιτική, αν θέλετε, και έτσι χάνονται δις ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι υπάρχει ε, πρόβλημα με την ε, ε, διαφυγή του κεφαλαίου από τη χώρα. Ξέρουμε ε, τι έγινε και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Ζούμε αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι οι συστάσεις αυτές βεβαίως φτάνουν αργά. Ένα μέρος όμως αυτών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να σταματήσουν οι καταχρήσεις οι οποίες, τις ε, και η κακή συμπεριφορά που υφίστανται κάποιοι μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είναι καλλιτυπίστοι σε κάποιες χώρες. Ξέρω ότι στην Ιταλία, στην περιοχή της Πούλια, υπάρχουν και κάποιοι μετανάστες που ήταν ε, εκ μέρους της μαφίας, έγιναν αντικείμενα και θύματα βίας και οι επιπτώσει πολλές φορές είναι τραγικές σε κάποιες Το δεύτερο ερώτημα τώρα. Το θέμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύη είναι μεγάλη σημασία τι θα κάνει η Ευρώπη. Στη συνθήκη εμφανίζεται η λέξη ε, αλληλεγγύη 20 φορέ. Και πολλές φορές οι όροι αυτοί εμφανίζονται ε, με πράξενο τρόπο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το άρθρο 222 της συνθήκης λέγει στα κράτη ότι θα πρέπει να επιδείξουν ελεγγύη εάν κάποια χώρα είναι θύμα ε, τρομοκρατικών ε, επιθέσεων ή φυσικών καταστροφών. Και εδώ γίνεται λόγος για επίθεση με χημικά ή με, με ε, πυρηνικά όπλα, αν υπάρξει σεισμός, καταποντισμός τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει το πρωτόκολλο το οποίο υπέγραψαν τα κράτη που λέει ότι οι συνθήκες της αλληλεγγύης θα πρέπει να καθιστούν από τα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι αλληλέγγυος με την ε, Κύπρο, αλλά στο πνεύμα. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα στην πράξη. Διότι ο καθένας αποφασίζει ε, à με μενού, όπως πάμε στο εστιατόριο, πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλληλεγγύη. Έτσι λοιπόν Τα πράγματα είναι έτσι ώστε όταν θα έχουμε ε, την σωστή ενημέρωση των πολιτών από άτομα όπως εσείς, θα μπορέσουμε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις. Πολλές φορές, ε, ακόμη και για θέματα γλωσσικής δυσκολίας δεν μπορεί κανείς να ζητήσει ούτε καν αυτά τα οποία μπορεί κάθε πολίτης να ζητήσει στη χώρα του. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, όπου έχουμε ε, πάντα πολύ περιορισμένες εξουσίες ε, ότι θα πάρουν τις αποφάσεις. Διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις διότι θα χρειαστεί για να τις εφαρμόσουν να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα. Ξέρουμε ότι πολλές χώρες δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το σύστημα λοιπόν αυτό ε, κινήτρων για τους ε, αξιωματούχους και τους ε, διπλωμάτες στο Συμβούλιο δεν θα αλλάξει παρά μόνο εάν υπάρχει πίεση εκ μέρους των πολιτών ε, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όσοι συμμετέχουν εδώ πέρα στις συζητήσεις και παίρνουν τις αποφάσεις, να έχουν μια προσέγγιση ευρωπαϊκή και όχι εθνική ο καθένας. και ελπίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται εδώ θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση στην Ευρώπη όπου θα μπορούμε να μιλούμε περισσότερο οι Ευρωπαίοι μαζί μας και να προτείνουμε και να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα. Εσείς, ε, ίσως ο καθένας στη χώρα του κάνει όσο σημαντική δουλειά κάνουμε και εμείς εδώ ο καθένας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Δύο μέλη έχουμε ακόμα για να δώσουμε το λόγο. Θα ήθελα να είστε σύντομοι γιατί έχουμε ακόμα δύο ερωτήσεις και στις 4.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Μπαργκέτσιο. η όλη η διαδικασία για την τράγκετα. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Η πρώτη δουλειά της τράγκετα είναι η εμπορία ανθρώπων σωστότατο. Αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι σε μεγάλο τμήμα της χώρας και της Ευρώπης η Ντράγκετα είναι η πιο ισχυρή εγκληματική οργάνωση και η οποία ασχολείται κυρίως με τη διακίνηση ναρκωτικών. Κανείς δεν θεωρεί ότι οι ταλέποροι πρόσφυγες είναι εμπόροι ναρκωτικών. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν μέτρα που δεν θα επιτρέπουν στη συγκεκριμένη οργάνωση να χρησιμοποιεί ε, πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες ή διαφόρους απελπισμένους για την ε, διακίνηση ναρκωτικών της και αυτό έχει ανακύψει από αρκετές έρευνες. Και για το θέμα αυτό θα έπρεπε και κατά την άποψή μου ότι είναι πολύ λογικό να επικρίνουμε τις διεθνείς οργανώσεις, όπως είναι καθόλου λογικό να επικρίνουμε και τους μισθούς των ευρωβουλευτών και πρέπει να πω ότι εγώ σε αντίθεση με κάποιους ε, ηθήνοντες ε, οργανώσεων ε, ήταν, ε, η στάση μου ήταν εναντίον ε, ηθινών των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως για παράδειγμα της ΦΑΟ και άλλων και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα στη διαστηριότητα της κυρίας του ΟΗΕ αλλά στη διαστηριότητα του ΦΑΟ που αποδείχθηκε ότι δαπανεί πολύ περισσότερα για τους υπαλλήλους της και για τους γραφειοκράτες της και πολύ λιγότερα για να μειώσει την πείνα στον κόσμο. Και από αυτή την άποψη εγώ θεωρώ ότι εάν θέλουμε να έχουμε σαφή νομοθεσία και με τη Eurodac ε, η δυνατότητα να ε, διαβιβάζονται στην αστυνομία δαχτυλικά αποτυπώματα είναι ένα θετικό βήμα κατά των ε, εγκληματικών δραστηριοτήτων, νομίζω ότι θα συνεισφέρουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ιερά δικαιώματα των ανθρώπων που πραγματικά δικαιούνται άσυλο και να δώσουμε την, πραγματικά, την πραγματική μάχη κατά της οργανωμένης μαφίας που είναι εχθρός του ανθρώπου και επομένως εχθρός ε, πρωτίστως των φτωχότερων και των πιο ευάλωτων όπως για παράδειγμα των μεταναστών και των ε, προσφύγων. Θα έπρεπε ορισμένες διεθνείς οργανώσεις να είχαν ε, θέσει το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων εναντίον αυτών των οργανώσεων και να μην θεωρηθεί ότι ε, πρέπει να δημοσιοποιείται αυτή η δραστηριότητα για να χρησιμοποιείται ως προεκλογική εκστρατεία. Ο κύριος Κρεταφυλίδης. Σύντομα, γιατί θα ήθελα να δοθεί μια επιπλέον ερώτηση. Ε, Θέλω να κάνω δύο μικρά σχόλια μόνο. Ε, νομίζω δεν απαντήσαμε στην εκπρόσωπο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ερώτηση ήταν... I want to... Ήθελα να πω ότι στην ερώτησή σας προηγουμένως εάν υπάρχει κανένα γραφείο το οποίο να αναλαμβάνει τους ε, ανήλικους μόλις... Το μικρόφωνο σα. Ε, αυτό που είπα είναι επειδή και η κυρία από τη Σουηδία επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και επειδή οι χώρε του Νότου, τουλάχιστον η Ελλάδα, η Κάζο και η Κύπρος έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί λοιπόν δεν φτιάχνουν γραφεία που να βοηθούν στη διαδικασία ασύλου ή μετεγκατάσταση ασυνείδητων, ε, ασυνόδευτων ανηλίκων ή άλλων ευάλωτων ομάδων. Διότι η Ελλάδα έχει απορριφθεί περίτρανα ότι δεν μπορεί να φτιάξει το σύστημα. Για να το φτιάξει θα υπάρξουν χρόνια και τα χρόνια σημαίνουν ακόμη περισσότερα θύματα και άνθρωποι που γυρνούν σαν σκιέ είτε στην Ελλάδα είτε εκτό Ελλάδα. Αυτό είπα γιατί δεν δείχνουν έμπρακτα και την παρούσα στιγμή την αλληλεγγύη τους με κάποιον άλλον τρόπο σύστημα αυτή τη στιγμή και αν μια χώρα όπως η Σουηδία μπορούσε να το κάνει θα ήταν ευχή έργο. Το άλλο το ζήτημα της γεωγραφικής ε, ε, διάστασης του ασύλου είναι γεγονός ότι υπάρχει ασχέτως ε, ε, εάν συμβεί κάτι, μια φυσική καταστροφή ή οπουδήποτε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι οι χώρε της Μεσογείου που δέχονται αυτά τα κύματα και επομένως το ζητούμενο είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος δίκαιης κατανομής των ευθυνών ανεξάρτητα από το ποια χώρα δέχεται τις πιέσεις αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. You have to... No, both. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Συγγνώμη. I would like Συγγνώμη. Έχουμε τέσσερα λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Όχι, όχι. Θα ακούσουμε και τις δύο ερωτήσεις. Και εσείς κυρία και η κυρία και μετά μια σύντομη απάντηση. Σύντομα όμως. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Greek. I Greek. Ε, θέλω μια διευκρίνηση. Λευτέρης Βιντέλλας από την εφημερίδα Έθνος. Ε, μια διευκρίνηση. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που περιμένουμε τον Μάρτιο, Απρίλιο, πότε θα έρθει τέλο πάντων, θα προβλέπεται η κατάργηση των κέντρων κράτηση προσφύγων, δηλαδή η Ελλάδα και όποια άλλη χώρα έχει τέτοια κέντρα, θα πρέπει να τα καταργήσει, θα πρέπει να κλείσουν όπω αναφέρθηκε η κυρία Βίκη Στρόμου πριν. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Ε, ε, και εσείς για την ερώτησή σας. Εκπροσωπώ το ε, πολωνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο και συγγνώμη για την ε, παρέμβασή μου. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται με το θέμα της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας ασύλου και έκλεισε το μικροφωνό της ομιλήτρια. Η κυρία Γουίκστρομ αναφέρθηκε ε, στη Λευκορωσία που είναι ένας από τους επικίνδυνους ε, γειτονές μας αλλά έχουμε πρόβλημα και εμείς ε, στα κέντρα κράτησης με την εκπαίδευση των παιδιών και ούτω καθεξής. Ο κύριος μας Επιντάλγο. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ. Καταρχάς να απαντήσω σε συγκεκριμένη ερώτηση για το αν κατά πόσο, και κατά πόσον από το Μάρτιο, Απρίλιο και μετά όταν πλέον θα έχει εγκριθεί η δέσμη μέτρων που σε μεγάλο βαθμό έχει εγκριθεί από τις κυβερνήσεις, μας λείπει ένα τελευταίο κομματάκι, γραφειοκρατικό, κοινοβουλευτικό εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ψηφίσουμε και εμείς στο Στρασβούργο, αν θα πρέπει να κλείσουν τα κέντρα κράτησης. Φυσικά, τα κέντρα κράτησης, τα οποία υπάρχουν στα σύνορα της Ευρώπης για πρόσφυγες, δεν εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία. Πρέπει να είναι ανοιχτά κέντρα και είναι ασύμβατο να υπάρχει ένα κοινό κρατούμενος με έναν ετώντα, ένα άτομο ο οποίος κάνει αίτηση ασύλου και υπάρχουν και μια σειρά από προϋποθέσεις που καθορίζονται στην οδηγία μας. Δεν είναι τόσο ακραία τα μέτρα όσο θα ήθελα εγώ ως εισηγητής. Ε, κάποιες κυβερνήσεις βέβαια θα ε, χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα ένα μεταβατικό διάστημα και θα χρησιμοποιήσουν και κάποια στιγμή την οποία θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν ε, τα παλιά σοφρονιστικά καταστήματα στις νέες ε, απαιτήσει ε, της νομοθεσίας η οποία θα τεθεί σε ισχύ. Βεβαίως και εμείς ως βουλευτές και εσείς ως δημοσιογράφοι και η κοινή γνώμη όμως πρέπει να επαγρυπνούμε και να φροντίσουμε να μην υπάρξει παρανομία σε αυτή την περίπτωση και να αποφύγουμε κάτι το οποίο είναι θεμελιώδη σημασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητά πολιτικό άσυλο δεν μπορεί να κρατείται. Αυτή είναι η βασική αρχή και από εκεί και πέρα μπορούμε να εξετάσουμε σε λεπτομέρεια κάθε ένα από τα θέματα. Κύριε Ταβάρες, στην ερώτηση της κυρίας από την Πολωνία για την κατάσταση με τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία. Eh, eh. Ακούστε. Η Πολωνία έχει εξωτερικά σύνορα, έχει τις υποχρεώσεις της εξαιτίας αυτού του γεγονότος όπως και τα άλλα κράτη-μέλη και στα πλαίσια του προγράμματος Frontex πρέπει να έχει και κάποια περισσότερα τεχνικά μέσα για να αντιμετωπίζει το θέμα της διαχείρισης των συνόρων, των εξωτερικών. Εκτός όμως από αυτή τη γενική παρατήρηση δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια άλλη ερώτηση, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. δεν θα καταλήξω σε συμπεράσματα, διότι δεν υπάρχουν ε, συμπεράσματα. Απλώς πρέπει να πω ότι μόλις τώρα άρχισε η συζήτηση επί αυτού του θέματος και έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά και σκληρή δουλειά. Ευχαριστώ τους πάντες. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και οι διερμηνείς σας ευχαριστούν, τους ε, ομιλητές και θα ήθελα να πω σε όλους τους δημοσιογράφους ότι όσοι από εσά θέλουν να κάνουν ε, την ε, οπτικοακουστική ε, επίσκεψη των εγκαταστάσεων, η Μπάρμπαρα Ροφ θα σας βοηθήσει, θα σας οδηγήσει στο άλλο κτίριο και όσοι θέλουν να επισκεφθούν το Παλαμεντάριουμ, το άλλο κτίριο, παραμείνετε έξω από την αίθουσα και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ε, ε, επίσκεψη, ε, ας μείνουν στην αίθουσα. Όσοι θέλουν να κάνουν και τα δύο, ας το κάνουμε τη σειρά. Ευχαριστώ πολύ σε όλες τις γλώσσες και χαίρετε.